Καλησπέρα σας. Θα προεδρεύσω στα ισπανικά. Bien, en primer lugar... Καταρχάς, μία ανακοίνωση από τις συνεδρίες των συντονιστών. Οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει αίτηση στη διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να διατυπωθεί προφορική ερώτηση με συζήτηση και ψήφισμα βάσει του άρθρου 36 και η αιτιολογία είναι διάσωση, έρευνα και διάσωση στην ε, ε, Μεσόγειο. Το κείμενο είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μεταξύ των εγγράφων ε, της ε, συνεδρίασης. Ε, σας το λέω πριν ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Είχαμε δύο πολύ έντονες ημέρες συνεδριάσεων και θα προσπαθήσουμε τώρα να προχωρήσουμε γρήγορα και σε αυτό το σκέλος συνεδρίασης Έχετε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να συνεισφέρετε σε αυτή τη συζήτηση. Στο σημείο 17 έχουμε την ακρόαση του υποψηφίου που επιλέγει για ε, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ, βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού. 2016-794 ε, και πρόκειται για τον κύριο Γιούρκεν Έμπνερ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτό το λέω και για τους καινούριους κυρίως, ε, η θητεία του παρόν εκτελεστικού διευθυντή ε, του κυρίου Μαρτίνου της Ευρωπέλ ε, πλησιάζει στο τέλος της, τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου του 2019. Η Ευρωπόλ δημοσίευσε την ανακοίνωση ε, για τη θέση στις 23 Ιανουαρίου του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ ε, υπέβαλε ένα κατάλογο περιορισμένο πέντε εξειδικευμένων επιρρογνωμόνων που ε, ενημέρωσαν το Κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο μάλλον αποφάσισε και ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι ο υποψήφιος είναι ο κύριος Έμπνερ στις 19 Ιουλίου. Στις 11 Ιουλίου οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν τον κύριο Έμπνερ βάσει των άρθρων 54 παράγραφος 2 και 55 παράγραφος 2 του κανονισμού της Ευρωπόλ. Τα άρθρα αυτά επιτρέπουν στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, ακούσει τον ε, υποψήφιο και ε, να γνωμοδοτήσει, αλλά η γνωμοδότηση θα είναι μη δεσμευτική. Κύριε Έμπνερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλώς ορίσατε. Προτείνω να ξεκινήσετε τώρα την παρουσίασή σας ε, για 10 με 15 λεπτά. Κατόπιν θα υπάρξει ε, μια διαδικασία ερωταποκρίσεων. Καλώς ορίσατε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας συστηθώ και να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου ως εκτελεστικού διευθυντή της Europol. Σκοπεύω να σας ε, παρουσιάσω και κάποια από τα προσόντα μου, διότι νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη της Europol. Πάντως ε, το πιο ενδιαφέρον για μένα θα ήταν να μάθω από σας ήδη σήμερα τι ερωτήσεις ε, έχετε εσείς για μένα ε, ή εμπασχευτώσει για τον μελλοντικό διευθύντη της Europol. Και βέβαια καθότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος, θεωρώ ότι σήμερα θα είναι μόλις η αρχή μιας συνεχιζόμενης συζήτησης. Μία από τις προτεραιότητές μου ως διευθυντή της Europol θα είναι να είμαι ε, και η επαφή για εσάς, ο εταίρος εσάς. Ε, γι' αυτό χαίρομαι πολύ για τη σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Όσον αφορά τα, προσω... τα επαγγελματικά μου προσόντα, θα ήθελα να αναφέρω ε, κάποια σημεία της ε, σταδιοδρομίας μου σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να κάνω και μια προσωπική παρατήρηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου να ε, θέσω υποψηφιότητα για την θέση αυτή. Πριν 34 χρόνια ξεκίνησα ε, στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας διότι με ενδιέφερε η δουλειά της αστυνομίας, με ενδιέφερε όμως και η διεθνή συνεργασία. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας είναι αρμόδια για την διεθνή συνεργασία ε, και αυτό ήταν ο βασικός λόγος που έκανα αίτηση εκεί. Όταν ολοκλήρωσα τον bachelor μου, ε, έγινα, ε, αξιωματικό προστασία προστασίας ε, υψηλών προσώπων, VIP. Γιατί αυτό έχει σχέση με τούτη τη θέση. Προσωπικά για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάστημα, διότι ήταν η εποχή επανένωση της Γερμανίας και βρέθηκα σε όλα τα ε, καυτά σημεία, στα σύνορα με την Ουγγαρία, με την Τσεχία, στα εσωτερικά σύνορα της Γερμανίας και για μένα Ε, το εσωτερικό σύνορο της Γερμανίας ήταν όχι μόνο προς την Ανατολική Γερμανία, ήταν και προς την Ανατολική Ευρώπη. Για μένα η Ευρώπη τελείωνε ε, στο σύνορο της Ανατολικής Γερμανίας ε, και για μένα ήταν η ιστορική η στιγμή που είχα την δυνατότητα να ζήσω την επανένωση όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και ε, της Ευρώπης όταν έπεσε το σιδηρούν παραπέδασμα. Διαπίστωσα δηλαδή τι ευκαιρίες ε, αλλά και κίνδυνοι συνδέονται με την ε, Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη λόγω των ιστορικών αυτών εξελίξεων. Όταν ήμουν αξιωματικό προστασία υψηλών προσώπων, είχα τη δυνατότητα να ε, σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο τη Βόνη, δημόσια διοίκηση και πολιτική οικονομία, διότι πάντα με ενδιαφέρει το οικονομικό έγκλημα. Για διάφορους λόγους όμως ε, τελικά δεν ε, κατέληξα ποτέ να διαρευνώ τέτοια εγκλήματα. Αλλά οι τεχνικές ε, προγραμματισμού ήταν πολύ χρήσιμες για μένα και στην αστυνομία, διότι οι αστυνομικές δυνάμεις σήμερα έχουν περιορισμούς όσον αφορά το δυναμικό. Γι' αυτό ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η θεωρητική γνώση. Κατόπιν ε, πέρασα στην ε, υπηρεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Ομοσπονδιακής ε, Γερμανίας. που λειτουργεί νυχτημερών και μια προσωπική παρατήρηση. Η σύζυγός μου τότε σπούδαζε ε, νομικά και ήθελε να γίνει δικαστής. Ε, πριν 25 χρόνια ε, άρχισα να εργάζομαι με χωρισμένο ωράριο, το 50% δηλαδή στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία και με μερική απασχόληση και το 50% στο σπίτι να φροντίζω το παιδί μας. Βέβαια πρέπει να οργανώσει κανείς τη δουλειά του, πρέπει όμως να λαμβάνει υπόψη και οικογενειακές πτυχές. Πρέπει να επιδιώκουμε και ισορροπία όσον αφορά τα δύο φύλλα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες που έχουμε. Αυτή λοιπόν ήταν μια χρήσιμη εμπειρία για μένα και ήταν χρήσιμη στη μελλοντική μου σταδιοδρομία. Είδα δηλαδή πώς πρέπει να συνδυάζει κανείς τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο αργότερα ε, ζήτησα να, ε, να πάω στην Αστυνομική Ακαδημία όπου ολοκλήρωσα το μάστερ μου. Το πρώτο ήταν πολιτική οικονομία, το δεύτερο έχει να κάνει με ε, τη δουλειά του αστυνομικού και ζήτησα τότε πρώτη φορά να πάω στη Europol. Υπήρχε τότε η δυνατότητα απόσπασης ως εθνικός εμπειρογνώμων και εργάστηκα για τον διευθυντή της Europol και ε, έκανα αίτηση ε, για να αναλάβω τη θέση του επικεφαλής ε, του γραφείου του διευθυντή της Europol και τελικά μου δόθηκε η θέση αυτή. Η Europol τότε ήταν πολύ καινούρια, όλα ήταν πολύ όμορφα, πολύ κομψά, όλα έπρεπε ε, να γίνουν από την αρχή, διότι ε, δεν ήταν ενσωματωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νομοθεσία και όλα αυτά έπρεπε να εκπονηθούν και Μα συζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol να αναπτύξουμε ένα σύστημα προγραμματισμού ε, και στρατηγικής και να ε, έχουμε περισσότερη λογοδοσία απέναντι στα κράτη-μέλη όσον αφορά τους πόρους που μας διαθέτουν. Ε, μου ανατέθηκε λοιπόν να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν το έκανα αυτό μόνος μου. Ε, αναζητήσαμε βέλτιστες πρακτικές. Ε, η ε, Αγγλία ήταν πολύ μπροστά τότε όσον αφορά αυτές τις στρατηγικές προγραμματισμού. Υιοθετήσαμε λοιπόν πολλές λύσεις που ήδη είχαν εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποια από τα θέματα αυτά. Θα τα συναντήσετε και σήμερα. Ε, για παράδειγμα, στις, εκθέσεις, ε, ε, στις εκθέσεις δραστηριοτήτων της Europol θα δείτε ότι βασίζονται στη δουλειά που είχαμε κάνει τότε. Ήμουνα και υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις και τότε κυρίως σε τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πολύ περιορισμένο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχε να πει κάτι, διότι ήταν πολύ περιορισμένες οι αρμοδιότητές του τότε. Ε, αυτό ε, επικρίθηκε επανειλημμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι αναζήτησαν επανειλημμένα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Europol. Κατόπιν έγινε αναπληρωτής διευθυντή της Europol, ήμουν αρμόδιο για, ε, για το ανθρώπινο δυναμικό και τα οικονομικά και πάλι για οικογενειακούς λόγους αλλά και για λόγους ε, επαγγελματική ε, σταδιοδρομίας αποφάσισα να αποχωρήσω νωρίτερα από τη θέση αυτή, διότι είχα μια καλή ευκαιρία πάλι στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, διότι δεν είχαν τότε εργαλεία στρατηγικής και προγραμματισμού και μου ζήτησαν λοιπόν να μεταφέρω τις εμπειρίες μου από την Europol ε, στο ΜΠΕΚΑ στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία για να εφαρμόσουν παρόμοιε λύσει. Μπόρεσα λοιπόν ε, τι ε, λύσει που είχαμε εφαρμόσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τι μεταφέρω και στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Και πρέπει να πω ότι νιώθω μια περηφάνεια. Το 2006 έγινε αυτό. Τώρα, ε, το 2019, χρησιμοποιούν ακόμα τα κεντρικά στοιχεία που είχαμε εφαρμόσει τότε. Επίσης, ήταν καθήκον μου να δημιουργήσω ένα δίκτυο για να έχουμε πιο στενή συνεργασία με ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις ε, ε, είχαν ανταλλαγές μαζί μας σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και είχα την δυνατότητα να συμμετέχω και σε αναλύσεις ε, διότι οι αστυνομικές δυνάμεις ε, δεν είναι απομονωμένες, ε, πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται στον κόσμο για να καθοριστούν οι ρυθμοί στο κάτω-κάτω του φορέα των αστυνομικών δυνάμεων. Μου ζητήθηκε να οργανώνω συναντήσεις όπως τον G7 ή επισκέψεις σημαντικών προσώπων από το εξωτερικό. Τώρα είμαι αρμόδιος ε, για την μονάδα κεντρικής, ε, ε, την κεντρική υπηρεσία πληροφοριών και έχουμε επαφές με τις επιχειρήσεις. Αναπτύσσουμε δηλαδή περαιτέρω το σύστημα πληροφόρησης Schengen, συλλέγουμε βιομετρικά στοιχεία για ταυτοποίηση και είμαστε το εθνικό σημείο επαφής για θέματα διαλειτουργικότητας και για όλων των ειδών ε, της αναζητήσεις. Αυτό είναι το βασικό μας ε, πεδίο ε, στην εργασία μας. Τώρα ζητώ να γίνω αναπληρωτής διευθυντής της Europol σε θέματα διακυβέρνησης. Αυτό έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, εξωτερικές σχέσεις, νομικές υποθέσεις και θέματα ασφάλειας. Έχοντας ακούσει την παρουσίασή μου, ε, ίσως αντιλαμβάνεστε ότι πολλές από τις ε, ε, από τη, ε, ότι μεγάλο μέρος των προσόντων μου συνδέεται και με αυτά που θα μου ζητηθούν στο μέλλον. Έχω δύο μάστερ, ε, έχω 20 χρόνια εμπειρίας εντός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, 10 χρόνια σε θέματα διακυβέρνησης, 7 χρόνια εμπειρίας σε, σε επιχειρήσεις και έχοντας εργαστεί 5 χρόνια στην Europol, νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω θετικά στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη της Europol. Πιθανές προτεραιότητες, ε, δηλαδή τι θα θεωρούσα εγώ σημαντικό. Ήδη αναφέρθηκα στο θέμα της διαχείρισης των πληροφοριών. Να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες της αστυνομίας από τη μία και ε, της προστασίας δεδομένων από την άλλη. Πρέπει η προστασία των δεδομένων ε, να ε, λαμβάνεται υπόψη ήδη από την αρχή σε όλες τις πτυχές εργασίας μας. Και βέβαια θα είναι καθήκον μου να στηρίζω τον Διευθυντή, θα είμαι ε, σύμβουλος, θα είμαι όμως και το σημείο επαφής για όλους τους εξωτερικούς φορείς, τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, αλλά και της ε, CEU που είναι πολύ ε, σημαντικό εταίρος της Europol. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα σημαντικό εταίρο και οι συνάδελφοί μου στη Europol λένε ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο για μα. Ε, μας υποστηρίζει και θα ήμουν ευγνώμων εάν ε, θα μπορώ να είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας ε, και να συμβάλλω και σε πολιτικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα ξεκινήσει ένα γύρο ε, συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε από του συντονιστέ μα καταρχά. Θα θέλαμε να περιορίσετε τι ερωτήσει σα σε τρία λεπτά και μετά ο υποψήφιος θα απαντήσει σε όλους στον πρώτο γύρο. Ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο εξ ε, του ΕΛΚ είναι η κυρία Πιτού. Η κυρία Ντυπών, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ήπνερ για την παρουσίασή σας. Ακούσαμε τις ε, γνώσεις ε, και την εμπειρία σας και προσφερθήκατε να διατηρήσετε τις ε, καλές ε, σχέσεις ανάμεσα στην Europol και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό στην πράξη πώς θα γίνει. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Και άλλο σχετικό θέμα. Πώς ε, θα είσαστε διαφανείς στην υποβολή εκθέσεών σας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Scrutiny Group, την ομάδα ελέγχου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είμαι και λίγο καινούργια με τα θέματα αυτά. Η κυρία Σίπελ, η οποία τα γνωρίζει, έχετε το λόγο, είστε συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Έμπνερ για την παρουσίασή σα και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχω την εντύπωση ότι δεν λέτε απλώ ότι σα αρέσει η ε, συνομιλία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το εννοείτε. Και σα διαβεβαιώ ότι θα επανέλθουμε από αυτού και ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για τι δύο πλευρέ. Επίσης, διάβασα όλα τα έγγραφα τα οποία μας στείλατε για τα προσόντα σας και μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο περιγράφετε τα επαγγελματικά σας προσόντα, αλλά και περιγράφετε και λίγο ε, πώς ε, συμβάλλει το πολιτικό περιβάλλον και η εμπειρία σας όταν μιλήσατε για την επανένωση της Γερμανίας, αλλά επίσης και τη σημασία της πτώσης του σιδηρού παραπετάσματος. Ε, όλες οι συζητήσεις που κάνουμε αυτές τις μέρες, ακόμα και στον τομέα της συνεργασίας με την αστυνομία, την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φαίνεται ή μπορεί και να ελοχεύει και ο κίνδυνος αυτός και δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάτι να πείτε από αυτού, ότι αυτές οι εξελίξεις σε κάποια από τα κράτη-μέλη μας όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία ή στην Πολωνία, που ήταν πολύ ευπρόσδεκτες στην αρχή και έγιναν πολύ καλές, καλά στην αρχή, ε, έκαναν πολύ καλά πράγματα ως ε, αρχικά μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης Στη συνέχεια η συνεργασία με αυτά έγινε πάρα πολύ δύσκολα. Ε, όχι ίσω στον τομέα τη αστυνομία, εσεί μπορεί να ξέρετε περισσότερα, αλλά σε θέματα δικαστική συνεργασία τουλάχιστον. Επίση, αναφερθήκατε και στο θέμα τη διαχείριση των πληροφοριών. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για το μέλλον, γιατί ο αριθμό των στοιχείων, ο αριθμό των πληροφοριών που συλλέγουμε ε, με τον ψηφιακό κόσμο που μα περιβάλλει θα αυξηθεί και αυξάνεται συνεχώ ε, και μάλιστα με δραματικό τρόπο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Εάν αφενό χρειαζόμαστε πληροφορίε, αλλά οι πληροφορίε που λαμβάνονται σήμερα είναι ήδη πάρα πολλέ. Είναι τόσο πολλέ και που χανόμαστε στο σύμπαν των πληροφοριών. Πιστεύετε ότι η ψηφιοποίηση ε, κάποια στιγμή εντό κάποιου χρονικού διαστήματο θα χρησιμεύσει προκειμένου να διαχωρίσουμε τι χρήσιμε πληροφορίε για εσά, για τη δουλειά σα στο αστυνομικό έργο με όλε εκείνε, οι οποίε είναι άχρηστε και απλώς συγχέουν και δημιουργούν πρόβλημα. Και πιστεύετε ταυτόχρονα χρησιμοποιώντα ψηφιακά μέτρα για τη διαχείριση όλων αυτών των πληροφοριών θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα ε, και επομένω τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σίπελ. Εξ ονόματο του Ρινιού υποθέτω ότι θα μιλήσει ο κύριο Τουντοράτσε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, συγχαρητήρια κύριε Έμπνερ που φτάσατε μέχρι εδώ και είστε ο υποψήφιος. Θα συνεχίσω με, από την τελευταία σας αποστολή. Μας είπατε ότι είσαστε ε, ε, διευθυντής τμήματος για τη διαχείριση των πληροφοριών. Μας είπατε ότι ε, έχετε εμπειρία από όσα γράφετε στο βιογραφικά όσα έχετε εργαστεί με βιομετρικά στοιχεία και διαλειτουργικότητα. Επομένω, η πρώτη με ερώτηση ε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τι άποψη έχετε εσείς προσωπικά, αλλά και ως ε, πιθανός μέλλον αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας που έχουμε τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια πιστεύετε ότι είναι τα ακριβή ωφέλη για την Ευρωπόλ από αυτό το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη σχέση σας με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Από όλα τα εργαλεία, κάποια από τα πιο καινοτόμα εργαλεία τα οποία έχει αναπτύξει η Ευρωπόλ ε, τα τελευταία χρόνια, πιστεύετε ότι αρκούν αυτά τα εργαλεία και είναι γνωστά επαρκώς από τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Πιστεύετε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη-μέλη και πιστεύετε ότι οι αστυνομικέ αρχέ στα κράτη-μέλη τα χρησιμοποιούν για του σκοπού και στο βαθμό ε, ε, για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί από τη Europol. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τουντοράτσο εξ ονόματος ε, του ID. Νομίζω εξ ονόματος της συντονίτρια, θα λάβει το λόγο ο κύριος Κόφορτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έπνερ που ήρθε εδώ σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του υποψηφίου και ε, έχω... Είχα τη χαρά να διαβάσω το βιογραφικό του κυρίου Έπνερ. Ε, δεν υπάρχει καμία αφιβολία, ε, Έχει πολύ πείρα. Έχω όμως μια ερώτηση. Διότι και στο βιογραφικό αλλά και στην παρουσίασή του ανέφερε τη δουλειά που έχει κάνει με το ΣΥΣ, το Eurodac και ε, είναι πολύ ε, ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά και σίγουρα θα δούμε πολλές εξελίξεις ε, τα επόμενα χρόνια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το τεχνολογικό δίλημα που έχουμε. Από τη μία δηλαδή, έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα στη δουλειά της αστυνομία. Με το CREST θα είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να μπορούμε να ε, μέχρι να μπορούν οι αστυνομικοί στον δρόμο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Από τη μία δηλαδή έχουμε δεδομένα τα οποία μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς αστυνομικούς σε όλη την Ευρώπη. Πώς ε, βλέπετε από τη μία το ότι έχουμε τόσες δυνατότητες με το δεδομένα, από την άλλη ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στους πολίτες όσον αφορά τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Έπνερ να μιλήσει για το δίλημα αυτό και πώς βλέπει τις εξελίξεις εντός της Europol τα επόμενα χρόνια. Εγώ Δανός είμαι, στη Δανία Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Europol ε, και η Δανέζικη αστυνομία θεωρεί ότι λειτουργεί καλά η σχέση αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Έπνερ ε, πώς βλέπει το δανέζικο μοντέλο ε, που εγώ βρίσκω ε, απόλυτα ικανοποιητικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόφο. το εξονόματος του ECR θα μιλήσει ο κύριος Ρίκο. Έχετε το λόγο. Señor Bricón. Señor Bricón. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Έμπνερ για την παρουσίαση. Ε, την παρουσίαση που μας κάνετε για την εμπειρία σας. Έχω μια ερώτηση για το μέλλον. Τι θέλετε να επιτύχετε ως αναπληρωτής εκτελεστικός διευθύντης της Ευρωπόλ. Ποιοι είναι οι στόχοι σας. Δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Δεν έχετε κάτι άλλο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Όχι μόνο αυτές, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρίβειά σας. Από την ΚΟΕ, η κυρία Ντάλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και Καλώς και ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Το θέμα ότι παρουσιάζεστε δημοσίως, είστε δημοσίως ε, για να πάρετε μια δουλειά σημαίνει ότι τη θέλετε πραγματικά οπότε και σίγουρα έχετε τα προσόντα. Ποιε είναι οι σκέψει σα όσον αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξη τη Ευρωπόλ ε, στο πλαίσιο των σημείων του σχεδίου του προγραμματικού εγγράφου. Μιλάμε για στρατηγικές προτεραιότητες ε, της Ευρωπόλ, όπως ε, παράδειγμα το να εξελιχθεί από έναν οργανισμό που βασίζεται σε, σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, σε μια ειδική η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ε, επιβολής του νόμου, δηλαδή από την επεξεργασία, από τη διεκπαιρέωση υποθέσεων να παράγει γνώση. Τι σημαίνει αυτό ρεαλιστικά, πιστεύω σημαίνει τη ε, ε των πληροφοριών ή το να πηγαίνεις σε άλλα μέρη για να βρίσκεις πληροφορίες, δηλαδή πας επιτόπου ε, η προτεραιότητα της Ευρωπόλ το να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιβολής του νομού, της έρευνας και της καινοτομίας. Και ποιοι θα είναι οι πιθανοί εταίροι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα σημαίνουν για σας συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και αν ναι, ποιο θα είναι το επίπεδο διακυβέρνησης σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας με δημόσιους φορείς. Ειδικότερα όσον αφορά τις αποστολές προσωπικού της Ευρωπολεκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ας πούμε για σκόπους συγκέντρωσης πληροφοριών. Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί αυτό. Φαντάζεστε να υπάρξουν περιπτώσεις να μην γίνεται αυτό μετά από αίτημα των αστυνομικών αρχών μιας τρίτης χώρας ή πώς θεωρείτε ότι θα διαμορφωθεί αυτό. Είμαι νέα στον τομέα αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ακριβώς τι γίνεται όταν στέλνουμε κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντάλη. Έχει ζητήσει επιπλέον το λόγο ο κύριος Ρος από το ECR. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Ρος. Ε, I just have the, the ECR ε, moment. So I have μιλώ εκ μέρους του ECR τώρα. Εγώ ρώτησα την ερώτησή μου ήδη όταν μίλησα εκ μέρους του ECR. Ωραία. Κύριε Θαρθαλό, εγώ έχετε εσεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έμπνερ, σα ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ ε, στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Είναι σαφές ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της αστυνομικής δουλειάς στο εγγύς μέλλον θα είναι η προσαρμογή σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο βιώνει τη νέα επανάσταση των νέων δικτύων, του 5G, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και θα ήθελα να ξέρω καταρχάς ποια είναι η αξιολόγησή σας ε, για την ε, προετοιμασία των αστυνομικών σωμάτων στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και δεύτερον, ε, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπόλ προκειμένου να ευνοήσει την προσαρμογή των αστυνομικών εργασιών σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρθαλέχος. Ο κύριος Σίκας από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπνέρη, για την ε, παρουσίασή σας. Ε, αναφερθήκατε στην προστασία των δεδομένων και ε, την ανάπτυξη των σχέσεων με το Κοινοβούλιο. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Και επίσης υπάρχουν ιδιαίτερα τμήματα του κανονισμού Europol που θα πρέπει να τροποποιηθούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Europol. Ωραία, και κλείνουμε το γύρο των παρεμβάσεων την, με την κυρία Φερικό ζητώ συγγνώμη και σας δίνω το λόγο. Μετά από αυτό θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Όμπνερ για να απαντήσει. Κυρία Μπρικμού. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Έμπνερ και συγχαρητήρια για την υποψηφιότητα σας. Έχω δύο ερωτήσεις κυρίω για εσάς. Η πρώτη αφορά τη συμφωνία συνεργασίας που έχουμε συνάψει με τρίτες χώρες. Ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες συνάπτονται με αυταρχικά καθεστώτα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι εχέγγυα μπορείτε να δώσετε ούτω ώστε να διαφυλάσσονται οι, αρχές, ε, οι θεμελιώδεις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, κάποιες υποχρεωτικές μελέτες επιπτώσεων είχαν διεξαχθεί για τη σύναψη υποχρεωτικά αυτών των συμφωνιών. Θέλω να μου πείτε την άποψή σα. Και μετά, για τα παιδιά, ο ρόλος τη Ευρωπούλη υπήρξε πολύ σημαντικό για την υλοποίηση Ευρωπαϊκή συνεργασίας ε, για την καταπολέμηση τη σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μεταξύ άλλων μέσω τη ταυτοποίηση των θυμάτων και την σύσταση μια task force. Ποιε είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον ε, της Αεροπόλ στο πλαίσιο αυτό και επιπλέον τι φιλοδοξία έχετε εσεί ω υποψήφιο για αυτή τη θέση στους τομεί που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και τι online εγκληματικέ δραστηριότητε κατά ανηλίκων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρικμόν. Κύριε Έμπνερ, έχετε τώρα τη δυνατότητα να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ε, έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε. So, 10 minutes of 10 λεπτά δεν είναι αρκετός χρόνος φυσικά για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, θα απαντήσω λίγο επιγραμμικά αν ε, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, ε, κύριε Αντιπό, ε, ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη σχέση ε, σε υψηλό επίπεδο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εγγυώμαι τη διαφάνεια. Η πρώτη μου απάντηση είναι η προσωπική μου παρουσία εδώ δείχνει ότι θα είμαι πάντα στη διάθεσή σα να απαντώ στι ερωτήσει σα και θα είμαι πάντα διαθέσιμος για οποιαδήποτε ερώτηση. Ωστόσο, Δεδομένου ότι είμαστε στι Βρυξέλλε, ε, είναι ευκολότερη η επικοινωνία. Αλλά όσον αφορά τα θέματα διαφάνεια, είναι σημαντικό να εκμεταλλευόμαστε όλε τι ευκαιρίε που μα δίνει ο κανονισμό ε, Ευρωπόλ. Ε, εκπρόσωποι του GPSG θα είναι επίση προσκεκλημένοι στι συναντήσει, οπότε και εσεί μπορείτε να έχετε συναντήσει ε, με την Ευρωπόλ. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να σα δίνουμε έγγραφα τη Ευρωπόλ. Το πιο σημαντικό είναι όσον αφορά την ετήσια, η ετήσια έκθεση επιδόσεων, μια γενική επισκόπηση των επιδόσεων τη Ευρωπόλ, θα μπορείτε να λαμβάνετε αυτό το έγγραφο, αλλά φυσικά θα έχετε και τη δυνατότητα να ζητήσετε και άλλα έγγραφα. Και από όσο ξέρω, πέρσι το Δεκέμβριο υπήρξε μια συνεννόηση εργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπόλ. Ούτω ώστε ε, έτσι έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε περισσότερε πληροφορίε από την Ευρωπόλ. Οπότε συνοπτικά, βάσει αυτών, ε, σα δίνω αυτή την απάντηση. Η κυρία Σίβελ ρώτησε για τις εξελίξεις στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Από άποψη αστυνομικού εξωματούχου μπορώ να σας πω ότι συμβάλλουν όπως και οι άλλες χώρες στις δεδομένων της Ευρωπόλ. Πρέπει να ακολουθούν το ίδιο καθεστώς υπό ποιε προποθέσει ε, συμβάλλουν, υπάρχουν κριτήρια ποιότητας και διασφάλιση που πρέπει να τηρούν. Οι διαστευρούμενοι έλεγχοι που κάνουμε βασιζόνται και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασία Δεδομένων, τον EDPS, τους Εθνικούς Επόπτες Προστασίας Δεδομένων που επίσης συνεργάζονται εκεί στο Συμβούλιο Συνεργασίας τη Ευρωπόλη. Υπάρχουν πολλά εχέγγυα λοιπόν για την επίβλεψη τη σωστή διαχείριση των πληροφοριών. Η διαχείριση των πληροφοριών τώρα είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε. Σχετίζεται με πολλέ ερωτήσει που ακούσαμε και με το ποιε είναι οι δυσκολίε ε, για την ε, Europol στο πλαίσιο τη διαχείριση πληροφοριών, το να βρει το σωστό ρόλο και το σωστό τρόπο αξιοποίηση των πληροφοριών. Το πρόβλημα τη Europol, όπω το έζησα εγώ εργαζόμενο στην Europol, είναι ότι ήταν πολύ λίγε οι πληροφορίε που λάμβανε η Ευρωπόλ. Ήταν, το πρόβλημα, το να δοθούν θα το θέμα είναι η Ευρωπόλ να λαμβάνει σωστέ πληροφορίε και σωστή ποιότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπόλ έπαιρνε πάρα πολλέ πληροφορίε. Κατακλυζόταν από πληροφορίε μόνο με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά μιλάμε για μια λειτουργία φιλτραρίσματο ουσιαστικά που φιλτράρει τις, ε, ε, που διαχωρίζει τι περιττέ πληροφορίε από τι πληροφορίε που είναι σημαντικέ για την αστυνομία. Αυτό θα βοηθήσει να, στην Ευρωπόλ να μπορέσει να αντιπροξέλθει στι δυσκολίε του μέλλοντο είναι κίνδυνος αλλά και ευκαιρία ταυτόχρονο η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει για καλύτερη προστασία των δεδομένων. Αν η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ε, δυνατό το να μην ασχολείται η αστυνομία με περτές πληροφορίε και αυτές τι πληροφορίε να έχουν εξαχθεί πριν ξεκινήσει η αστυνομία μια έρευνα, έτσι συμβάλλει ενεργά στην προστασία των δεδομένων. Όσον αφορά ναι, την ερώτηση για τα βιομετρικά στοιχεία και το πλαίσιο διελειτουργικότητας και ποια θα είναι τα ωφέλη για την Ευρωπόλ. Η ατζέντα διελειτουργικότητας σε όλο το φάσμα αφορά την αρχιτεκτονική στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Ευρωπόλ. Αυτό είναι σημαντικό. Αν μπήκαν σε περισσότερε λεπτομέρειες, η Ευρωπόλ θα έχει τη δυνατότητα και ήδη το μελετά ε, στο πλαίσιο του SIS. Η Ευρωπόλ θα παίξει σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά πληροφορίε που σχετίζονται με την ασφάλεια, ε, που σχετίζονται με την προστασία των συνόρων, τη εξέλιξη τη μόλις ε, υιοθετηθούν τα σχετικά έγγραφα και η Ευρωπόλ επίσης και αυτό είναι το σημαντικότερο, θα είναι ο φορέα όπου οι αστυνομικέ δυνάμει από ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν υπό όρου να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων τη μέσω μία interface ενία. Δεν θα χρειάζεται πλέον να έχει κανεί πρόσβαση σε κάθε βάση δεδομένων ε, υποβάλλοντα ξεχωριστή αίτηση. Εφόσον έχει κανεί τα δεδομένα, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων και να ψάχνει πράγματα με ένα κλικ σε όλε τι σχετικέ βάσει δεδομένων και να βρίσκει τουλάχιστον ένα hit. Οπότε θα αξίζει τον κόπο. Αυτό όσον αφορά την ατζέντα διαλειτουργικότητα, πολύ σημαντικό και για την Ευρωπόλ. Όσον αφορά τι σχέσει με τα κράτη-μέλη, και εσεί κάνατε αυτή την ερώτηση, όταν γνωρίζουν τα εργαλεία, ε, ε, ε, ναι, οι απαιτήσει των κρατών μελών είναι περισσότερε από ό,τι μπορεί να παρασχεί η Ευρωπόλ αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει σχέση και με τον προπολογισμό που συζητήσατε πιθανότατα και χθε και σήμερα το πρωί. Ένα από τα ζητήματα όπου η Ευρωπόλ θα μπορούσε να παίξει σημαντικότερο ρόλο και στο μέλλον θα ήταν να προσφέρει ε, πλατφόρμες συνεργασία όσον αφορά το κυβερνό έγκλημα. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τι ίδιε ανάγκε ε, να έχουν πλατφόρμες αποκρυπτογράφηση ε, αποκωδικοποίησης για να μπορούν να διερευνούν ε, έγκλημα, ε, κυβερνοεγκλήματα στο μέλλον. Θα είναι λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμο το να υπάρχουν σε ένα κεντρικό σημείο μια τέτοια πλατφόρμα. Απομένει πολλή δουλειά να γίνει και σε αυτό το τομέα και στις επικοινωνίε και για περαιτέρω ε, πρόθεση της Ευρωπόλ, για περαιτέρω αξιοποίηση της Ευρωπόλ. Αν δείτε την έκθεση ετήσιας δραστηριότητας, αν δείτε τα νούμερα πέρυσι, δείχνουν πολύ θετικά σημάδια. Πάνω από 4 εκατομμύρια έρευνε γίναν ε, πέρυσι στο σύστημα πληροφοριών τη Ευρωπόλ. Πάνω από ένα εκατομμύριο μηνύματα κυκλοφόρησαν μέσω των διάβλων Σιένα. Αυτό δείχνει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται περισσότερο από ποτέ. Αλλά φυσικά υπάρχει και περιθώριο ανάπτυξη. Ο Ευρωβουλευτής από τη Δανία ρώτησε αν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό δίλημα μεταξύ αφενός των δυνατοτήτων χρήσης των πληροφορικών συστημάτων αφετέρου ταυτόχρονα τηρώντας ε, τα εχέγγυα ε, απορρίτου. Θα έλεγα ότι δεδομένων των νέων ε, συστημάτων προστασία των πληροφοριών που έχουμε, νομοθετημάτων για την προστασία των πληροφοριών, έχουμε αυτέ τι δυνατότητε. Από την αρχή μπορεί κανεί να εισάγει, αναπτύσσοντα μια υποδομή πληροφορική, από το σχεδιασμό μπορεί να προβλέψει προστασία δεδομένων, να εισάγει απαιτήσει από την αρχή όπως εργάζονται σήμερα τεχνολογικά συστήματα, τα συστήματα πληροφοριών, ε, βασίζονται όχι μόνο στις βάσεις δεδομένων, αλλά και στους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται. Οπότε έχουμε εκεί ατομικά δικαιώματα πρόσβαση και μπορούμε να παρακολουθούμε περισσότερο την προστασία των δεδομένων και να επαληθεύουμε ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που είχε προβλεφθεί. Ο ε, κύριο Ρο, ε, ρώτησε για του στόχου. Εγώ ω αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή τη Ευρωπόλ Του έχω στην περιγραφή της δουλειά μου. Είναι να υποστηρίζω τη διευθυντή. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η διευθύντρια. Πρέπει να τη βοηθώ και να διαχειρίζομαι ε, τις δραστηριότητες. Ε, σε σχέση με αυτή τη δουλειά φυσικά άλλοι στόχοι ε, το είπα και στην αρχική μου παρουσίαση θεωρώ ότι θα μπορούσα να εξέλιξω περισσότερο τη διαχείριση πληροφοριών στην Ευρωπόλ γιατί δεν σχετίζεται μόνο με την πληροφορική έχει να κάνει και με ε, διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και αυτός θα είναι ο στόχος μου με περιορισμένο προπολογισμό δεν θα είναι εύκολο έχουμε και περιορισμένη στελέχωση οπότε θα πρέπει να οριστούν οι σωστές προτεραιότητε και να στελεχωθούν ανάλογα και μετά θα δούμε πώς θα ε, εξελίσσονται οι επιδόσεις μέσα στα χρόνια ένα από τα ζητήματα που δεν ανέφερα πιστεύω από τα σημαντικότερα είναι το να ε, είσαι συντονιστής ασφάλειας της Ευρωπόλ το να μεριμνάς για το προσωπικό για την ουσία και για τις πληροφορίες που διαχειρίζεται η Ευρωπόλ. Στρατηγικές προτεραιότητες μόλις τις ανέφερα, καινοτομία και έρευνα. Με ρώτησαν κατά πόσο μπορεί να χρειαστεί συνεργασία με ιδιώτες. Με τον ιδιωτικό τομέα, ναι, σίγουρα. Ε, στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος είναι αδύνατο να γίνει χωρίς συνεργασία με τους ε, παρόχους ε, υπηρεσιών online, ε, με τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ. Και εκεί υπάρχει μια διάκριση μεταξύ του τι επιτρέπεται στο πλαίσιο της εντολής Ευρωπόλ, στον κανονισμό της Ευρωπόλ, όσον αφορά την εκπαιρέωση δεδομένων με ιδιώτες. Αυτό δεν προβλέπεται, αλλά με τη χρήση τεχνολογικών που, που έχουν αναπτύξει ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να μας βοηθήσουν στο μέλλον. Η αστυνομία δεν μπορεί να προγραμματίσει Παντό είδου προγράμματα και εφαρμογές από μόνη τη, θα χρειαστεί να αποκτήσει ε, προγράμματα από ε, τρίτα μέρη που θα παρέχουν ωστόσο τα χέρια τα οποία απαιτούνται για τις αστυνομικέ δραστηριότητες. Συγκέντρωση πληροφοριών για τρίτες χώρες ε, και η συνεργασία με τρίτες χώρες αναφέρθηκε από κάποιον άλλον. Ο κανονισμό τη Ευρωπόλ το λέει καθαρά. Η Ευρωπόλ από μόνη τη δεν μπορεί να διαπραγματευτεί συμφωνίες ε, συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια γι' αυτό ε, μαζί με το Συμβούλιο. Τέτοιου είδου διαπραγματεύσει γίνονται βάσει ιεραρχία. Το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπόλ είναι ότι μπορεί να συνάψει ε, συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες περιορισμένες στην ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών και μη προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί κίνδυνος μια τρίτη χώρα να μην τηρήσει τα ζητήματα προστασίας δεδομένων της ε, Ευρωπόλ ε, κατά την πρόσβασή της ε, βάσης δεδομένων της Ευρωπόλ. Οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτη χώρα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα τίθεται η ερώτηση της, του κατά πόσο είναι επαρκές το σύστημα προστασίας δεδομένων που έχει αυτή η χώρα με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα είναι αδύνατο να συναυθεί συμφωνία συνεργασίας οι ψηφιακές εξελίξεις, ε, μόλις αναφέραμε 5G, τεχνητή νοημοσύνη, την ανέφερα, το 5G θα είναι δύσκολο για την αστυνομία, το ακούσατε και χθε. Θα πρέπει να προσέξουμε, σεβόμενοι φυσικά τα δικαιώματα του πολίτη και την ανάγκη για απόρριτο, αφενός αφετέρου πρέπει και η αστυνομία να μπορεί να κάνει τη δουλειά στο μέλλον. Στο σημερινό επίπεδο του 5G η αστυνομία δεν είναι δυνατόν να ε, εντοπίσει ε, τις απαραίτητες προφορίες στο μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν το απόρριτο, αλλά θα πρέπει κάπως να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μια από τις μεγάλες δυσκολίες ε, που ανέφερα θα είναι η ψηφιοποίηση. Με ρωτήσετε ποιε είναι οι μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις και αν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι στον κανονισμό της Ευρωπόλου. Δεν είμαι νομικός. Φυσικά έχω μελετήσει τον κανονισμό της Ευρωπόλ ε, προετοιμαζόμενος για αυτή τη θέση και ξέρω ότι μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα εδώ και εκεί όπου μπορεί να ε, χρειαστεί να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ένα από τα ζητήματα, για παράδειγμα, που συνάντησα εγώ ε, αφορά τη συνεργασία με ιδιώτες που τώρα ε, διοχετεύεται στις ομάδες, στις εθνικές ομάδες διαχείρισης της Ευρωπόλ, αλλά αυτό πρέπει να το αναθεωρήσουμε ενδεχομένω. είναι θέμα νομοθέτη. Αν γίνει αναθεώρηση του κανονισμού τη Ευρωπόλ, φυσικά η Ευρωπόλ μπορεί να συμβουλέψει βάσει τη δική της εμπειρία και μετά ο νομοθέτη αποφασίζει τι είδου τροπολογίε τροποποίηση θεωρεί ότι είναι απαραίτητε. Συγγνώμη, ξέχασα τι μπορεί να γίνει με την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την εμπορία ανθρώπων. Έχετε δίκιο. Και τα δύο αυτά θέματα αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπόλ. Όχι μόνο εμπορία ανθρώπων, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα ή παράνομη μετανάστευση που δεν στρεφόμαστε κατά των μεταναστών αλλά κατά των εγκληματικών δικτύων που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους ε, και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών. Ακολουθώντας τον κύκλο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτά τα τρία ζητήματα ανήκουν στις τρεις προτεραιότητες της Ευρωπόλ, όπου εξορισμού η Ευρωπόλ συμμετέχει μέσω στρατηγικής ανάλυσης. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, βάσει επιχειρησιακή ανάλυση, αλλά και με ενεργέ έρευνε υποστηρικτικέ, με ερευνητικέ ομάδε, αλλά και με την παροχή οικονομική ε, επιχειρησιακή βοήθεια και με έρευνε που γίνονται από τι ε, δημόσιε αρχέ και το καθεξής. Αυτά είχα να πω ως απαντήσει στις ερωτήσεις που ακούσαμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Έμπνερ για τις πολύ συγκεκριμένε και εκτεταμένες εξηγήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους. Πρέπει να προτείνω τώρα την συνέχεια της διαδικασίας για τα επόμενα βήματα αυτής της ακρόασης. Επειδή επήγει η γνωμοδότηση, πρέπει να αποσταλεί στο Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να επιλέξουμε τον υποψήφιο και να ξεκινήσει ο διορισμός του τον Οκτώβριο η γνωμοδότηση πρέπει να σταλεί στον πρόεδρο όλοι ε, ως πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και η πρόταση της Προεδρίας Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι να σταλεί πρόταση στους συντονιστές ε, για έγκριση, για να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη σου, ε, για να κάνουν που θεωρούν ότι χρειάζονται σήμερα. Και στις 6 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο σχολιασμός ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τον πρόεδρο της γνωμοδότησης ε, για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για την άποψη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ε, εάν ε, δεν υπάρχουν ενστάσεις μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι λοιπόν μετά από την ακρόαση που κάναμε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις Μέχρι τις 4 η ώρα θα διακόψουμε ακριβώς και θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Καθίστε παρακαλώ. Πρόκειται για το σημείο 18. Θα ακούσουμε την παρουσίαση των ε, καθηκόντων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από το Διευθυντή της, τον Μάικολ Φλάχερτη. Όπως γνωρίζετε, ιδίω ε, όσοι από εσά ε, έχετε εμπειρία σε αυτή την επιτροπή, ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ω εντολή να παρέχει στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε με ίδια πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διάρκεια των ετών, η κατοπιν αιτηματος του ευρωπαικου κοινοβουλιου στη διαρκεια των ετων η επιτροπη ΛΥΜΠΕ ε, έχει μόνιμη συνεργασία με τον οργανισμό και ο οποίο οργανισμό παρήχε εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε πολλού τομεί και απάντησε στα αιτήματα γνωμοδότηση που ζήτησε η Επιτροπή ε, που αφορούσαν διάφορες νομοθετικές προτάσεις. Ε, ευχαριστώ τον Μάικολ Φλάχερτη ο οποίος ε, πάντα είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να μας παρουσιάσει τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του οργανισμού στα νέα μέλη και την καλή συνεργασία που είχαμε ανέκαθεν μαζί του. Είναι πάντα χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας. Έχετε το λόγο, έχετε 15 λεπτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για το θερμό καλωσόρισμα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ μπροστά σας. Όπως είπε και η Πρόεδρος πολύ καλύτερα από μένα, η σχέση μεταξύ μας ε, είναι στενή, ισχυρή σχέση και για μας είναι η πιο σημαντική σχέση που έχουμε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, στην Επιτροπή για τον ιστορικό ρόλο για την προώθηση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου, γιατί δύσκολα έχω αυτή την ευκαιρία να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τη Γραμματεία που είναι φίλος της, ε, του οργανισμού. Ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, τα βασικά ε, θα σα πω για εισαγωγή. Ο βασικό μα ρόλο είναι να στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν λέω θεσμικά όργανα, αναφέρομαι φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη. Ο ρόλο μα λοιπόν δεν είναι ρόλο πολιτική, δεν είναι εκτελεστικό, δεν είναι λήψη αποφάσεων. Είναι ε, συμβουλευτικό ε, και υποστηρικτικό. Είναι ουσιαστικά τεχνικό ρόλο. Έχει σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρησιμοποιώ και εμένα τον όρο, διότι φυσικά αναφερόμαστε μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα όπω περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σχετίζονται και με την Ευρωπαϊκή Αρμοδιότητα. Δεν είμαστε ένα γενικό οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή σύνθεση. Ε, αντικείμενό μας ε, επίσης ε, τα θέματα που μας αποσχολούν ε, δίνονται κυρίως από μια σειρά από θέματα τα οποία μας δίνονται από καιρούς καιρούν το πολιετές πλαίσιο. Το πολιετές πλαίσιο την χάνει διαπραγμάτευσες μεταξύ των συνομοθετών και καθορίζει σε αδρές γραμμές κάποιους θεματικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Όχι σε όλους γιατί μπορούμε να πάμε και πέραν του πολιετούς πλαισίου ιδίω όταν αναλαμβάνουμε ένα αίτημα από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Και το δικό σα το θεσμικό όργανο, το Κοινοβούλιο, μέσω τη Επιτροπή, ήταν ε, αυτό ο οποίο ε, συνήθω απευθύνει αιτήματα προ εμά ε, για τομεί τη εντολή μα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και εκτό του πολιετού πλαισίου. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο ε, εργαλείο, μια πολύ πλούσια εργαλειοθήκη, την οποία χρησιμοποιήσαμε για τη δουλειά σας. Θα τα αναφέρω και θα σας δώσω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το πρόγραμμα εργασίας σας. Έρευνες, καταρχάς. Τα Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κάνω τις πιο φιλόδοξες και πολύ συχνά παγκοσμίω μοναδικές έρευνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την άποψη του κατόχου του δικαιώματος. Ζητάμε τους δικαιούχου ε, για διάφορα ζητήματα. Τι εμπειρία έχουν προκειμένου εσείς, οι πολιτικοί πολιτικοί ηθήνοντε να ανταποκριθείτε στι ανάγκε και στα προβλήματά σα. Θα σα δώσω παραδείγματα για όλα εντό ολίγου. Δεύτερον, μαζί με τη συλλογή δεδομένων μέσω τη διαδικασία των ερευνών που είναι ποσοτική, κάνουμε και ποιοτική έρευνα. Ε, παραδοσιακή εφαρμοσμένη έρευνα για το τι έχει αποτελέσματα και τι όχι ε, στα θέματα που μα απασχολούν στη κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερα επίση ότι εργαζόμαστε σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα στοιχείο τη δουλειά μα, το οποίο θα περιμένατε φυσικά και είναι και ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι στο βαθμό που έχει σημασία. Ε, δημιουργούμε συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών. Σπανίως επιλέγουμε την τάδε ή τη βίνα χώρα. Λέμε ότι ε, το θέμα μπορεί να αντιμετωπίζεται ή δεν αντιμετωπίζεται με συγκριτικό τρόπο ε, σε όσα κράτη-μέλη έχουν σημασία από αυτού. Επίσης γίνονται και εκθέσεις για συγκεκριμένα ε, ζητήματα ε, περιοδικά. Είναι πολύ ε, δύσκολο να τα εξηγήσω αυτά σε δύο λεπτά. Έχω δύο πράγματα όμως ακόμα πριν σας δώσω παραδείγματα. Το επόμενο είναι ο οργανισμό πλέον δραστηριοποιείται τόπου. κάτι το οποίο θα εκπλήξει αυτού που μα γνωρίζουν και χρόνια. Δεν είμαστε θεωρητικοί οι οποίοι καθόμαστε στα γραφεία μα. είμαστε εκεί έξω και ασχολούμαστε με θέματα στα οποία έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Μπορεί να είναι δημιουργία ικανοτήτων, μπορεί να υποστηρίζουμε με κάποιο τρόπο τους ανθρώπους τόπου. προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε τη διαφορά. Και φυσικά ε, υπάρχει κάτι το οποίο θα αναφέρω και ω παράδειγμα σε ελίγου. Ε, στη διάρκεια ζωή του οργανισμού εκτιμούμε ε, ότι έχουμε τη δυνατότητα να συγκαλέσουμε κόσμο, να συνενώσουμε ανθρώπους για να γίνει η απαραίτητη δέσμευση ώστε να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα. Τώρα, να σας τα παρουσιάσω όσοι έχουν στην πραγματικότητα, τους τομείς εργασίας που ενδιαφέρουν εσάς. Ο πρώτος είναι η μετανάστευση. Η μετανάστευση ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στην κορυφή ε, το, ε, ε, των προτεραιοτήτων. Ε, οπουδήποτε υπάρχει το θέμα, ε, ασχολούμαστε με το θέμα. Φέτος το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή ε, στα ε, μοντέλα θανάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Είδαμε τι γίνεται, παρακολουθήσαμε ε, τις διαδικασίες και στα δικαστήρια και επιστήσαμε την προσοχή και στα αποτελέσματα των αποφάσεων. Όταν φτάνει κάποιο στις ακτές, δεσμευόμαστε στα σημεία υποδοχής, τα λεγόμενα hot spots και εκεί υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία με την ΕΑΣΟ, με τη Frontex και με τους άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς που ασχολούνται με τα θέματα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν. Σε μεγάλο βαθμό ασχολούμαστε και με την ε, προστασία των παιδιών και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και τις δυνατότητές τους ε, να ανταποκριθούν σε σεξουαλική βία. Ε, και όταν λέω τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, εννοώ τα πάντα. Από συμβουλές, ε, από το να υπάρχει φωτισμός ε, στα κέντρα υποδοχής, πού θα μπουν αυτά τα φώτα, πώς μπορούμε να φερόμαστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια κτλ. Παρακολουθούμε τους μετανάστευση σε όλη τη διαδικασία μετανάστευσης μέχρι την επιτυχία ή την αποτυχία της ένταξής τους. Και εδώ γίνεται και ποιοτική έρευνα, καθώς και έρευνες για να μπορέσουμε χαρτογραφήσουμε τις εμπειρίες αυτές. Και τέλος, στον τομέα τη μετανάστευση, και αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο κάνουμε περιοδικέ ε, δημόσιες εκθέσεις, ε, κάνουμε λεπτομερείς ε, δημόσιες εκθέσεις κάθε τρει μήνες για την κατάσταση στις, στα κράτη-μέλη που πλήττονται περισσότερο. Αυτό θεωρείται ότι είναι μία αξιόπιστη πηγή εις βάθος πληροφοριών για το θέμα αυτών, από 15 έως 17 κράτη-μέλη. Ο δεύτερος τομέας, στον οποίο θα σας παρουσιάσω ως παράδειγμα, είναι ο τομέας της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα τομέα όπου υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη δέσμευση από τον οργανισμό μας, ε, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε αιτήματα τα οποία έχουμε λάβει από εσά. Για παράδειγμα, ε, βάσει ενός αιτήματός σας ε, πριν από κάποια χρόνια, υπήρξαν ε, πολύ λεπτομερείς ε, ε, διαδικασίες εξέτασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών είναι η συνήθις ποιοτική έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη και σας δίνουμε τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε εσείς τη δουλειά σας. Επίσης, μας ζητήσατε και μας ενθαρρύνατε να προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, μέσω της ανάπτυξης ε, μεγάλων βάσεων δεδομένων στα ευρωπαϊκά σύνορα από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς η Επιτροπή σας ε, λάβατε υπόψη πολλά από τα στοιχεία τα οποία σας προτείναμε στα αποτελέσματα τα οποία σας ε, ε, παρουσιάσαμε. Ε, η ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων έχει πολύ στενή σχέση με το πολύ λεπτό ζήτημα της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων, τη δυνατότητα να ε, συνομιλούν μεταξύ τους. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό, χάρη σε εσά, είναι κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα ε, γιατί λαμβάνεται υπόψη και τις προτάσεις μας και την ανάλυση μας. Και τέλος, στον τομέα αυτό θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεσμευόμαστε ακράδαντα και είμαστε πάρα πολύ αποσχολημένοι με το θέμα της χαρτογράφησης των θεμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Προσφάτως, για παράδειγμα, δημοσίευσαμε δύο εκθέσεις στο πλαίσιο αυτό, μία πάρα πολύ πρόσφατα, τις προηγούμενες εβδομάδες, ε, για τα λεγόμενα ε, dirty data, πώς ε, ε, προβλήματα ε, δημιουργούνται στη ζωή μας όταν είναι λανθασμένα, είναι προϊόν διάκρισης και δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό και ακριβώς ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ασχολείται με θέματα τεχνικής νοημοσύνης. Τρίτον και τελευταίο, ως παράδειγμα της δουλειάς μας, είναι το, ο τομέας της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Εδώ έρχομαι στις έρευνές μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τις έρευνές μας και γνωρίζουμε από την απάντησή σας σε εμά είναι ίσως το πιο χρήσιμο υλικό το οποίο σας δίνουμε, ε, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Βία κατά των γυναικών το οποίο σε μεγάλο βαθμό ήταν κάτι το οποίο ε, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα χάρη στην έρευνά μας για το θέμα αυτό πριν από 7 χρόνια. Ακόμα δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη δουλειά. Οι Εβραίοι στην Ευρώπη, η δική τους εμπειρία. Πέρσι δημοσιεύσαμε τα απορίσματά μας και μάλιστα τα παρουσιάσαμε και εδώ στην Επιτροπή για το τι σημαίνει να είναι κανείς Εβραίος στην Ευρώπη σήμερα, κάτι το οποίο δημιούργησε ευρύτερη συζήτηση και μια υπενθύμηση του πώς οι έρευνες αυτές μπορούν να οδηγήσουν και τη δέσμευση από πλευρά πολιτική. που χρειάζεται. Ε, ε μειονότητες στην Ευρώπη, κυρίως ε, ε, μετανάστες μειονοτήτων, η Ρωμά που μας αποσχολούν και δύο άλλα πράγματα τα οποία είναι προσεχή. Στο τέλος του έτους θα δημοσιεύσουμε τη δεύτερη έρευνα και τα πορίσματά μας για το τι σημαίνει να είναι κανείς ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 120 άτομα απάντησαν στη διαδικτυακή έρευνα 120.000, ε, δεν ήθελα να πω 120, συγγνώμη, 120.000 άτομα απάντησαν στη διαδικτυακή μας έρευνα και μπορώ να σας, δεν μπορώ να σας παρουσιάσω ακόμα τα πορίσματα γιατί είναι σε διαδικασία επεξεργασίας, αλλά είναι παραδοσιακός τρόπος συνεργασίας μαζί σας. Θα σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα εάν θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα. Και η δεύτερη προσεχής μας έρευνα, που είναι η τελευταία που αναφέρω ως παράδειγμα, είναι ότι στο τέλος του έτους και στις αρχές του 2020 θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας ε, ε, έρευνας που έγινε για πρώτη φορά παγκοσμίω. Ε, μια έρευνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μια έρευνα για τη στάση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ ε, πουθενά αλλού. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά προσβλέπω στην παρουσίασή τους εδώ σε εσά. Πριν ολοκληρώσω, τι ακριβώς κάνουμε μαζί σας. Ε, πολλές τρόπους έχουμε αναπτύξει. Μου λένε εδώ να μιλάω λίγο πιο αργά. Μιλάω σε Ιρλανδούς όλη μέρα, επομένως ε, ε, αντί να προσέχω να μιλάω αργά αγγλικά, ε, το πέταξα από το παράθυρο και έβαλα πέμπτη ταχύτητα, ζητώ συγγνώμη. Μιλάμε λοιπόν μαζί σας ε, συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όταν μας προσκαλείτε για να σας πούμε τα πορίσματά μας, να σας παρουσιάσουμε τις ερευνές μας, να σας παρουσιάσουμε τις εκθέσεις μας σε θέματα που σας ενδιαφέρουν, είμαστε πάντα έτοιμοι να έρθουμε να το κάνουμε. Ε, ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμη αυτή η συνεργασία, αλλά δεν είναι μόνο η επίσημη συνεργασία. Είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε διαθέσιμοι και συνολικά αλλά και ατομικά ως ε, πηγή, ως πόρος πληροφοριών. Έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα και αναλύσεις από όσα χρειάζονται και παρουσιάζονται στις εκθέσεις και στα ε, έρευνε μας και θέλουμε εδώ να σας τα παρουσιάσουμε. Είμαστε στην υπηρεσία σας. Κάθε μέλος της Επιτροπής αλλά και η ίδια η Επιτροπή μπορεί να αποτανθεί σε εμά για να τους ε, πούμε τα πορίσματά μας. Τρίτον, Συνεχίζουμε να είμαστε ε, διατεθειμένοι να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, ε, είτε ε, για ποιοτική έρευνα, είτε για χνομοδοτήσεις, για ευαίσθητα θέματα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είχαμε την πρώτη έκθεση, για παράδειγμα, για τα hot spots κατόπιν αιτήματό σα ή και για την εκπόνηση νομοθεσία. Μπορούμε να σα δώσουμε μια πιο νομική ανάλυση ενό σχεδίου νόμου. Επίσης, σας καλούμε να συμμετέχετε και στις δικές μας εκδηλώσεις, εάν θεωρείτε ότι είναι πολύτιμο. Κάθε τρία χρόνια φιλοξενούμε την πιο ουσιαστική συζήτηση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, που λέγεται το Φόρουμ των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γίνεται στη Βιέννη. Η επόμενη θα γίνει το 2021. Η ΛΥΜΠΕ πάντα στέλνει ισχυρέ αντιπροσωπείε, οι οποίε διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο του Φόρουμ των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Επίση, ελπίζουμε ότι θα μα επισκεφτείτε στη Βιέννη. Η πάγια πρακτική μα είναι να καλωσορίζουμε οποιαδήποτε φυσικά επίσημη αποστολή προ εμά που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί, αλλά θα θέλαμε να σα αναφέρουμε και ότι η πόρτα μα είναι πάντα ανοιχτή, όχι μόνο κάθε τρία χρόνια, Οποιαδήποτε ευκαιρία λοιπόν να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τι κάνουμε και να εργαστούμε πρακτικά για να σε υποστηρίξουμε είναι ε, ευπρόσδεκτη. Για να ολοκληρώσω, τα βασικά ανέφερα τη Βιέννη. Η έδρα μας είναι στη Βιέννη. Είμαστε περίπου 105 άτομα. Ε, αλλά αν συμπεριλάβετε και τις άλλες κατηγορίες ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας στο κτίριό μας, είμαστε περίπου 150 άτομα. Ο πλήρης προϋπολογισμός μας το 2019 είναι 22.500.000, αλλά από αυτά μόνο τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ είναι ο επιχειρησιακό προϋπολογισμός μας. Όλα όσα σας περιέγραψα και πολλά από αυτά που δεν ανέφερα προσπαθούμε να τα κάνουμε λοιπόν με 6,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν είναι φυσικά ε, παρά μία σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προσβλέπω στη συζήτηση κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φλάχερτη. Δεν ε, αμφιβάλλω ότι θα υπάρχει πολύ σημαντική ε, εκπροσώπηση από πλευράς ΛΥΜΠΕ στο θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στους ε, βουλευτές. Και καταρχάς, η κυρία Γιάροκα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chair. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Καθώς και που έρχεστε στην ΛΥΜΠΕ κάθε τόσο για να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολλές πληροφορίες που μας δώσατε. Δύο ερωτήσεις έχω για θέματα που αναφέρατε εν μέρη ή καθόλου. Σήμερα το πρωί είχαμε τον κύριο Τίμερσμαν εδώ στην αίθουσα που μιλούσε για το νέο μηχανισμό για ένα κράτος δικαίου και ως ανθρωπολόγος ε, τον ρώτησα πώς βλέπει τη μεθοδολογία ενός τέτοιου μηχανισμού δεδομένου ότι πολλά από τα εργαλεία που έχουμε, τουλάχιστον στο χαρτί, για να ε, καταπολεμούμε τις παραβιάσεις του, του κράτους δικαίου υπάρχουν, δεν χρησιμοποιούνται όμως πολλά από τα ωραία πράγματα που κάνετε δεν χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ στο παρελθόν είχαμε και διπλά μέτρα και σταθμά και γι' αυτό μερικές φορές τα κράτη-μέλη θυμώνουν για την κατάσταση αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας σε θέματα όπως είναι τη φτώχειας των Ρωμά ε, και λοιπά. Ε, σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε εσείς και οι συνεργάτες σας τα τελευταία 15 χρόνια καθώς και που μας βοηθήσατε να, ε, να εκπονήσουμε την στρατηγική για τους Ρωμά. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η μεγαλύτερη έλλειψη είναι, και το γνωρίζετε επειδή εσείς έχετε τα δεδομένα ε, στα χέρια σας, ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη καλής παρακολούθησης. Γνωρίζω ότι υπάρχει τεχνογνωσία στο γραφείο σας. Ε, οι συνεργάτες σας μου εξήγησαν ότι ο κρίκος που λείπει είναι η επιτόπου έρευνες ε, με τις ομάδες στόχους ε, αυτές καθ' αυτές. Θα στηρίξετε λοιπόν την Επιτροπή μας ε, στην προσπάθεια να έχουμε ένα πρόγραμμα 3 εκατομμυρίων ευρώ για να εφαρμόσουμε προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάροκα. Σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να μιλάτε λίγο λιγότερο και να προσπαθήσετε να μιλάτε ένα-δυο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σπούρεκ. Ε, thank you, madam. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, παρουσίασή σας. Ε, ως ε, αναπληρώτρια επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, της Πολωνίας ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τώρα ασχολούμαι με την προσχώρηση στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την βία εις βάρος των γυναικών. Καταλαβαίνω ότι μια σειρά κρατών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ένα πιλωτικό πρόγραμμα συλλογής δεδομένων ε, το 2018 και 2019 μέχρι να προχωρήσουν στην κανονική συλλογή δεδομένων το 2020-2021. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποια ήταν αυτά τα πιλωτικά κράτη, ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής τους ε, και πώς έχει αναπτυχθεί η μεθοδολογία για την έρευνα αυτή και θα ήθελα επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τα Άτομα ΛΟΑΤΚΙ που ξεκίνησε ο οργανισμός σας φέτος τον Μάιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα τελικά συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα το 2020. Ήθελα να ρωτήσω όμως αν υπάρχουν κάποια προκατακτικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ την κυρία Σπούρη και κυρία Νταλή. Okay. Señora Dalí, usted la palabra. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας ε, και προσλέπω στην καλή συνεργασία με τον οργανισμό σας. Έχω ακούσει μόνο καλά λόγια Νομίζω ότι οι έρευνε ε, που κάνετε για να λαμβάνονται περιστατημένε αποφάσεις είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές. Θα ήθελα να ρωτήσω, σας ζητήθηκε γνωμοδότηση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά το Brexit και τι συνέπειες του Brexit στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα γνωρίζετε ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με διαδικασίες απέλασης ε, και Υπάρχουν ανησυχίε για τα άτομα που, για παράδειγμα, ε, αυτή τη στιγμή αποτελούν ε, αντικείμενο ε, ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Μετά το Brexit οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν χωρίς προστασία και υπάρχει η σύμβαση του 1957 για τις απελάσεις και εκδόσεις, αλλά δεν δεν παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε προηγούμενο ε, κράτους μέλους που γίνεται τρίτη χώρα. Τι θα γίνει λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές, ε, τι θα γίνει για τους ανθρώπους που δεν ε, θα προστατεύονται πια από το, από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σας έχει ζητηθεί να εκπονήσετε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό ε, ή πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και ω Ευρωβουλευτής, πώ μπορεί να σας προσεγγίσει κανείς ε, για να λάβει γνωμοδότηση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Κούνκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κυρία Διευθύντα. Ω πρώην υπουργό Δημοκρατίας της Σουηδικής Κυβέρνησης είχα την ε, δυνατότητα να εξετάσω τη δουλειά σα και χρησιμοποίησα εκθέσεις σας για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, Σουηδική πολιτική. Με ανησύχησε όμως τότε και ακόμη με ανησυχεί η δυνατότητα του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων ε, να μας ε, διαβιβάζει δεδομένα και γεγονότα, διότι αναφέρατε τον περιορισμένο προϋπολογισμό σας. Ως διευθυντής ε, είστε το πρόσωπο με την καλύτερη γνώση των όσων δεν μπορείτε να κάνετε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε παραδείγματα πραγμάτων που δεν μπορείτε να κάνετε, που πιστεύετε όμως ότι είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Σήμερα το πρωί είχαμε συζήτηση με τον κύριο Τίμερμανς για το κράτος ε, δικαίου και καταλαβαίνω ότι η δουλειά του οργανισμού σας στόχο έχει την προστασία των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Πριν ε, δύο εβδομάδες, Γάλλος αστυνομικός αποκάλυψε ότι 500 Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μπει σε μαύρη λίστα. Μπορεί λοιπόν να παρεμποδιστεί η ελεύθερη τους κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά με αφορμή την ε, Σύνοδο Κορυφής ε, του Μπιάριτς. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν εσείς γνωρίζετε την ύπαρξη τέτοιας μαύρης λίστας και ποια θα ήταν η προσέγγισή σας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ενετφέλτ. Και έχουμε έναν ακόμα ομιλητή πριν απαντήσει ο κύριος Φλάχερ. Κύριε Φλάχερτη, σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά που κάνετε. Νομίζω ότι δεν εκτιμάται επαρκώς ε, δημοσίως η δουλειά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχω μια ερώτηση ή παρατήρηση. Η κυρία Λίβια Γιάροκα είπε νωρίτερα ότι Ε, πολύ συχνά ε, τα κράτη-μέλη ή μάλλον οι κυβερνήσεις δυσανασχετούν με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, τομέα θεμελιωτών δικαιωμάτων. Κάποιοι άλλοι μπορεί να επικροτούν την τις ενέργειες αυτές. Εσείς λοιπόν εξετάζετε περιπτώσεις διακρίσεων, ρητορικής μίσους και έχουμε την τάση να εξετάζουμε συγκεκριμένες ε, ομάδες της κοινωνίας ε, που ε, το κάνουν αυτό. Υπάρχουν όμως πολιτικά κόμματα, υπάρχουν θρησκευτικές ομάδες που επίσης έχουν ρητορική μίσους και παρακινούν ανθρώπους στο μίσος και θα ήθελα να ρωτήσω, νιώθετε ότι έχετε εσείς την ελευθερία να επικρίνετε τέτοιες ομάδες ε, και είσαστε διατεθειμένος να εξετάσετε ε, το πώς η ρητορική μίσους από ε, αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων και πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν την ρητορική μίσους εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ακόμα μιλητέ. Ζήτησε κάποιο ακόμα το λόγο και με αυτό κλείνουμε τον ε, κατάλογο των αγορητών. κυρία Στρίκ. Like Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάχερτη για την ε, δουλειά που έχει κάνει και να τον συγχαρώ για την ε, δουλειά του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Χρησιμοποιώ τα αποτελέσματα των εργασιών σας και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Ε, ε, ε, ενεργείτε συμπληρωματικά σε σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης. συνεργάζεστε μαζί τους και αν το συγκρίνεται με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φαίνεται να έχουν κάπως ε, ευρύτερο πεδίο εργασίας. Ε, έχουν ε, παρεμβάσεις τρίτων, παρέχουν συμβουλές στα κράτη-μέλη, καλούν κυβερνήσεις να κάνουν κάποια πράγματα ή να αποφύγουν κάποια άλλα. Και η κυρία Κούν και η κυρία Ινετφέλτ αναφέρθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις. Νιώθετε ότι η εντολή σας είναι αρκετά ευρεία ώστε να είναι αποτελεσματική ε, για να μπορέσετε να αλλάξετε κάποιες πολιτικές και πρακτικές. Και τέλος ε, θα ήθελα να μιλήσω για το εύρος θεμάτων με τα οποία ασχολείστε. Μιλήσατε για πολιτικές ε, μετανάστευσης, την εξωτερική διάσταση της πολιτικής μετανάστευσης. Τι κάνει ο οργανισμός σας στο θέμα αυτό. Θεωρείτε ότι αρκεί η εντολή σας για να μπείτε και σε αυτόν τον τομέα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα κλείσουμε με δύο ακόμα αγορητές. Ο κύριος Βαντεντρίσε. Σωστά, σωστά το είπατε. Ευχαριστώ. Τρέκα zoals gewoonlijk. Ehm, heel interessante uiteenzetting. Eh, bedankt daarvoor. Μια χαρά το zijn op cijfers en niet op σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ πέρα. Έχω εξετάσει τις, ε, ε, ε, τα έντυπα που έχετε εκδώσει, για παράδειγμα, για την Ισλαμοφοβία. Φαίνεται να υπάρχει και αύξηση του αντισημιτισμού. Έχουμε μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Κάποια κράτη-μέλη υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με την εθνοτική καταγωγή των ε, ε, εγκληματιών και των θυμάτων. Ε, στο Βέλγιο δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, στις κάτω χώρες όμως ναι και στη Γερμανία ναι. Υπάρχει επισκόπηση των δεδομένων αυτών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το προφίλ των εγκληματιών. Ωραία. Και για να κλείσει ο γύρος των παρεμβάσεων των Ευρωβουλευτών, η κυρία Κάνκο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ε, δεν άκουσα όλη την παρουσίαση σας, ε, διότι ε, κατέφθασα κάπως αργά. Έχω μια ερώτηση όμως για τα δικαιώματα των γυναικών, διότι Ε, και στο παρελθόν ε, έχω εξετάσει τις εκθέσεις σας. Ε, έλεγε μία από αυτές ότι το 1 τρίτο των γυναικών πέφτουν θύματα βίας, λεκτικής σωματικής, το 1 πέμπτο είναι θέματα stalking. Και Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα δεδομένα αυτά για μας. Ε, μπορείτε να μιλήσετε λίγο για την ε, Eurostat και για την ε, ομάδα που εργάστηκε σε θέματα της βίας με βάση το φύλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε λοιπόν 10 λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιάρακο, ε, εσείς ρωτήσετε την πρώτη ερώτηση για τα εργαλεία, για το κράτος δικαίου και το βαθμό στον οποίο ενδεχομένως υπάρχουν αλλά ε, υποχρησιμοποιούνται. Ε, μια από τις δυσκολίες είναι να βρει κανεί αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των 28 κρατών μελών που υπογραμμίζουν την ύπαρξη μηχανισμών που υπονομεύουν το κράτος δικαίου αναγνωρίζουμε και εμείς ότι είναι σημαντικά αυτά τα αποδεδεικτικά στοιχεία. Τα δεδομένα της ΦΡΑ συγκεντρώνονται από τη ΦΡΑ. Δεν ξέρω αν τα ανέφερε ο κ. Τίμερμαν σήμερα το πρωί, αλλά στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου αναφερόμαστε στο σύστημα πληροφοριών για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη, όπου συγκεντρώνουμε οτιδήποτε υπάρχει ω στοιχείο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλου του οργανισμού, με σκοπό να βοηθούμε εσά και όλου του υπόλοιπου ε, που θα διαχειριστείτε μηχανισμούς σημερινούς και μελλοντικού ε, στη δουλειά σας. Αναφέρθηκε το ζήτημα των Ρωμά. οι εργασίε για τα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτό στις του πληθυσμού δεν έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι απογοητευτικό και συμφωνώ μαζί σα. Η αποτελεσματική παρακολούθηση με συνέπειε είναι κάτι που θα μπορούσε ακόμα να ενισχυθεί. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και την αιρεσιμότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή τι χρήματα θα δοθούν εκεί ε, πώς θα δαπανηθούν μάλιστα τα κονδύλια αυτά. Θεωρούμε ότι έχουμε ενθαρρυντικά σημάδια. Συζητείτε να δοθούν σε οργανισμούς, εθνικούς οργανισμούς θεμελιδών δικαιωμάτων και ισότητας περισσότερα κονδύλια σε εθνικό επίπεδο για να ε, δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε αυτό στους κλάδους. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα για να φέρει αποτελέσματα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αναφέρατε, κύριε Γιωρεκά, Δημερώσω, ενδεχομένω αν θέλετε στείλτε μου περαιτέρω πληροφορίε, γιατί δεν είμαι επαρκώ πληροφορημένος για να σα δώσω μια σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή. Κύριε Μπούρεκ, ρωτήσατε ε, για την βία κατά των γυναικών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση τη. Ήταν πριν να ε, αναλάβω εγώ τη θέση μου, θα ζητήσω από του συναδέλφου μου να σα στείλουν τι πληροφορίε, γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να σα δώσω μια πλήρη απάντηση τώρα. Ωστόσο, μπορώ να απαντήσω για του ε, ΛΟΑΤΜΕ. Ε, και τη σχετική έρευνα. Τα πρώτα ευρήματα θα έρθουν του χρόνου, αλλά περιμένουμε και κάποια αρχικά ευρήματα φέτο, του επόμενου μήνε, πριν κλείσει το έτο. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Κυρία Ντάλη, ε, για την ερώτηση που κάνατε. Δεν έχουμε ασχοληθεί μέχρι στιγμή ε, να αναλύσουμε τι συνέπειε του Brexit σε θέματα θεμελιδών δικαιωμάτων. Θα ξεκινήσω μάλλον από κάπου αλλού. Όπω φαντάζεστε, και εμένα με ενδιαφέρει το ζήτημα προσωπικά δεν θα το ξέρετε εγώ υπήρξα ε, ε επίτροπος ε, για την Επιτροπή Βορειοϊρλανδίας, οπότε γνωρίζω το θέμα σωστά. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε εμπλακεί διότι ένα οργανισμό σαν το δικό μα ήταν σημαντικό να μην περιπλέξει τη διαπραγμάτευση περαιτέρω. Αλλά την κατάλληλη στιγμή, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για έναν οργανισμό σαν εμά να συμμετέχει ε, ρεαλιστικά, θα είμαστε έτοιμοι. Δεν κάνουμε τέτοια έτοιμη διότι δεν εντάσσεται στου δικού μα τομεί αρμοδιοτήτων, αλλά αν μα ζητηθεί και είναι η σωστή στιγμή και δεν πρόκειται να προκαλέσουμε περισσότερε επιπλοκέ, είμαστε έτοιμοι. Κυρία Κάνκε, θέσατε το ζήτημα του προπολογισμού και το σε ποιο βαθμό ο προπολογισμό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, απαντώντα. Ε, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε νέου τομεί εργασία, να κάνουμε ελέγχου διακριτική μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο, τον έχει αναπτύξει σε παγκόσμιο επίπεδο να εξετάσουμε τι επαγγελματικέ πρακτικέ ε, ε, στο χώρο εργασία, να δούμε τι διακριτική μεταχείριση υπάρχει ενεργό με το πώ είναι το πρόσωπό σου, τι εθνικότητα είσαι, πώ επηρεάζει αυτό το αν βρίσκει δουλειά. Ε, υπάρχουν έλεγχοι διακριτική μεταχείριση, είναι ακριβή ε, κοστίζουν πολύ, αλλά δεν έχουμε, και δεν έχουμε τους πόρους εμείς για να ξεκινήσουμε τέτοιες έρευνες. Και μετά στους τομείς που ήδη δραστηριοποιούμαστε μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα των όσων κάνουμε, αλλά υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε ακόμα ε, κάνει. Στην Ελλάδα έχουμε έναν άνθρωπο, φανταστείτε. Είναι απογοητευτικά και στέλνουμε ανθρώπους από τη Βιέννη. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο. Ναι, καλά πράγματα κάνουμε, αλλά χρειαζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ε, είχαμε ανθρώπους ε, στη Μόρια, στο ε, καταβλισμό αυτή τη βδομάδα, αλλά πρέπει να επισκεφτόμαστε διαρκώ όλα αυτά τα hot spot, όλα αυτά τα κέντρα υποδοχή. Όχι μία φορά μόνο. Και είναι αδύνατο γιατί δεν έχουμε πόρου. Περικόπτουμε τον προπολογισμό μα από όπου μπορούμε για να μπορέσουμε να τον παρουσιάσουμε στο Συμβουλίο μα. Είναι πολύ σκληρό, ξέρετε, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Παίρνουμε ένα συγκεκριμένο κλάδο όπου γίνεται πολύ καλή έρευνα, για παράδειγμα ανάπηροι άνθρωποι που έρχονται να ζήσουν ε, κάπου και κάνουμε πολύ καλή έρευνα και μετά λένε οι συνάδελφοι ας πάμε τώρα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να φέρουν αποτελέσματα αλλά δεν έχουμε χλεφτά. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει κάτι που δεν κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Κάτι άλλο να σας πω για τον προϋπολογισμό. Οι συνομοθέτες τα θεσμικά όργανα αυξάνουν διαρκώ τον προπολογισμό οργανισμών με πολύ ευαίσθητε λειτουργίε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ASO, Frontex, του λέτε όλο και περισσότερο να κάνουν τη δουλειά του με τρόπο που να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και μετά στρέφονται σε εμά για βοήθεια, για να φέρουν τα αποτελέσματα που προσδοκείτε εσεί, αλλά εμεί δεν έχουμε του επιπλέον πόρου. Του λένε δηλαδή, «Ε, κάποιοι παίρνουν έξτρα συνοριοφύλακε και εγώ δεν μπορώ να πάρω το ένα έξτρα άτομο που χρειάζομαι. Ανέκαθεν είχαμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα, αλλά ξέρετε, χρειαζόμαστε και του συνομοθέτε με το πλευρό μα. να αναγνωρίσουν ότι το σκληρότερο, όσο σκληρότερα γίνονται τα πράγματα στι κοινωνίε μα, τόσο μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται και τόσο περισσότερη δουλειά έχει ο οργανισμός μας. Ε, κύριε Μπρενερα, ε, συγγνώμη που δεν προφέρω καλά το όνομά σας δεν ασχολούμαστε με επιμέρους περιπτώσεις, με συγκεκριμένες υποθέσεις ε, ε, καταχρήσεων και παραβιάσεων. Δεν έχουμε τις δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να καταγράψουμε ζητήματα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και να τα αναφέρουμε σε εσά, στον κόσμο, μέσω της ετήσιας έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, παρέλειψα να την αναφέρω νωρίτερα. Παρουσιάζουμε τέτοια, σα υποβάλλουμε τέτοια έκθεση κάθε, κάθε χρόνο όπου καταγράφονται διάφορα ζητήματα, αλλά φυσικά πρέπει να είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πάει στραβά στι κοινωνίε δεν, είναι πάντα, δεν εντάσσεται πάντα στην αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πεδίο αρμοδιοτήτων. Κυρία Νέτφελτ, με ρωτήσατε αν φοβόμαστε να επικρίνουμε κυβερνήσει. Όχι. Αν θέλουμε να δούμε καταχρηστικέ ε, πρακτικές ηγετών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα το κάνουμε ήδη. Δείτε, ε, δεν ντρεπόμαστε, κατονομάζουμε ακόμη και το λόγο μίσου, οποιασδήποτε περιπτώσει όπου διακρίνουμε προβλήματα. Το πρόβλημα του λόγου μίσου στην Ευρώπη έχει οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που οι ηγέτε τη βγάζουν καθαρή. Ναι, ε, στο πλαίσιο της εντολή μα, ε, τη λειτουργία μας, των ικανοτήτων που έχουμε, δεν φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα όπω έχουν. Ε, ε, κύριε Στρίκ, ε, ρωτήστε για τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ένα από τα ζητήματα όπου ένας άνθρωπος σαν εμένα λέει «Πολύ χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί έχει σημασία». Αν δεν είχαμε φανταστική συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν θα τα καταφέρναμε πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής. Είναι συμπληρωματικό το έργο μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Καταρχάς είχαμε διαφορετικές λειτουργίες Εμεί δεν λαμβάνουμε αποφάσει ε, που μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν, ενώ το δικαστήριο μπορεί. Έχουμε διαφορετικέ θητείε, δηλαδή διαφορετική εντολή. Δεύτερον, συναντιόμαστε πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, για να ευθυγραμμίζουμε, να συντονίζουμε τι εργασίε μα, ούτω ώστε να επιτυγχάνονται αυτέ οι αρχέ που ανέφερα. Υπάρχει πάντα εκπρόσωπο του Συμβουλίου τη Ευρώπη στο Συμβούλιο μα. Αυτό είναι ασυνήθιστο για οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και εγώ έχω προσωπικά σχέση με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ασθενέ ε, σχέσει ε, και πολύ καλέ. Ε, το Συμβούλιο τη Ευρώπη έχει ευρύτερη εντολή από εμά και φυσικά είναι αυτό. Ωστόσο, εμεί δεν είμαστε ο μόνο οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Έχουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντολή για θεμελιώδη δικαιώματα, για να το πω έτσι. Και εσεί. Δεν είμαστε οι μόνοι, λοιπόν. Ε, που ασχολούμαστε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πάντα φυσικά μπορούμε να διευρύνουμε την εντολή μα, να τη βελτιώσουμε. Το Συμβουλίο μα το ζητά διαρκώ. Αυτή είναι η γενική μου απάντηση. Ένα θέμα που θέλω να σα επισημάνω όσον αφορά την εντολή είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα δεν συναδεί με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιδών Δικαιωμάτων η δική μα εντολή. Αυτό είναι λίγο παράξενο και πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εμεί μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με θέματα αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μόνο εφόσον μα το ζητήσουν τα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι πολύ περίεργο για ε, έναν οργανισμό, για μια δομή που ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω εμεί. Θα θέλαμε στο μέλλον να μα δοθεί μια ευκαιρία να αναθεωρηθεί τεχνικά η εντολή μα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Με ρώτησαν επίση, ε, εσεί νομίζω, κυρία Στρέκ, για την εξωτερική διάσταση τη μεταναστευτική πολιτική. Εκεί έχω να σα πω ότι εκεί μπορούμε μόνο να κοιτάξουμε τι εξωτερικέ δραστηριότητε των θεσμικών οργάνων ή των κρατών μελών. Δεν μα επιτρέπεται βάσει τη εντολή μα να εξετάζουμε τι δράσει ε, τρίτων κρατών. Ο κ. Βεντεντρίσε ε, ρώτησε για διάφορα ζητήματα, για τα θύματα κατάχρησης ε, και επιθέσεων, να ψάχνουμε να βρούμε τους ε, υπεύθυνου ε, και φυσικά ναι ψάχνουμε, αλλά οι απαντήσεις είναι πολλές και διαφορετικές. Και έγινε και μια ερώτηση για τη μετανάστευση. Ξέρετε, πρέπει να καταπολεμήσουμε όλους τους μύθους που έχουν γεννηθεί για τη μετανάστευση. Λένε ότι οι μετανάστες έχουν φέρει τη σεξουαλική βία στην Ευρώπη δεν είναι αλήθεια. Ήταν δικό μα το πρόβλημα και υπήρχε πολύ καιρό πριν του μετανάστε. Το γεγονό ότι μια πράξη σεξουαλική βία διαπράττει από έναν μετανάστη δεν είναι το ίδιο σαν να λε ότι οι μετανάστε έφεραν τη σεξουαλική βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν κάθε φορά που, γεννιούνται, που παρατηρούμε τέτοιου μύθου είναι αβάσιμοι. Ε, δεν τεκμηριώνονται από τίποτα. Και τέλο η τελική ερώτηση από την κυρία Κάνου ε, για διάφορα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών δεσμευόμαστε για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ε, στο πλαίσιο και της ε, διαφορετικής μεταχείρισης των φύλων. Δεν υπάρχει μία έρευνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα που να μην περιλαμβάνει μια ειδική διάσταση για τις γυναίκες. Είναι στάντρα διαδικασία πια για μας. Ε, Όπως παρουσίασα και στην Επιτροπή σας πέρυσι, είχαμε συγκεκριμένο κομμάτι της έκθεσης για τις γυναίκες Ρωμά, για τις μετα... γυναίκες μετανάστες. Μετά, όσον αφορά την Eurostat και την προετοιμασία για την επερχόμενη έρευνα για τη βία κατά των γυναικών, δεν έχω στα χέρια μου τις λεπτομέρειες, αλλά δεσμεύομαι να, σας τα, στείλ, να τα στείλω στην κυρία Κάνκο αυτέ τι πληροφορίε δήμερος πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο. Ήταν εξαιρετική συζήτηση και ελπίζουμε να σας δούμε πολύ σύντομα. Και φυσικά ε, η Επιτροπή μας που πάντα είναι σε επαφή με τον οργανισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί συναδέλφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η παρουσίαση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων των ε, Ευρωπαίου Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων. Θα γίνει από τον κύριο... Βιεβιορόσκι. Βιεβιορόσκι ο οποίος είναι ε, αναπληρωτής επόπτης. Θα του δώσουμε απευθεία το λόγο για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε προσκαλέσει ε, τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Είναι τιμή να ε, εμφανίζομαι εδώ τόσο σύντομα μετά τις εκλογές. Από την άλλη, ε, θα ευχόμουν να μην είμαι εδώ σήμερα, διότι αντικαθιστώ τον αγαπητό μου φίλο, τον κύριο Πταρέλη, τον οποίον ε, χάσαμε πριν δύο εβδομάδες. Ο Τζοβάνι Εκτιμούσα ιδιαίτερα την Επιτροπή σας ε, και τα μέλη και τα μέλη της ε, και ήταν ε, αμοιβαία τα αισθήματα. Όσοι τον γνώριζαν καλά, συγκινήθηκαν από την τιμή που του κάνατε χθες το πρωί. Ο πρόωρος ε, χαμός του Τζοβάνι ήταν θλιβερός, αλλά το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τις ε, εργασίες του τα τελευταία δέκα χρόνια αρχικά ως ε, αναπληρωτής επόπτης και κατόπιν ως επόπτης προστασίας δεδομένων. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω σύντομα τον ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ε, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και η προστασία των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποτελούν αντικείμενο εγγράφων που σας έχουμε στείλει και ηλεκτρονικά και που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ο ε, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι ανεξάρτητος και εξετάζει τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι ε, οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τα, προσωπικά δεδομένα, τον ιδιωτικό βίο και να, προωθήσουμε, να προάγουμε τις καλές πρακτικές στα 67 θεσμικά όργανα και οργανισμούς που εποπτεύουμε ιδιαίτερα καθήκον, τα συγκεκριμένα καθήκοντά μας αναφέρονται στο στον κανονισμό 2018 σε 1725 και κάποιες άλλες νομικές πράξεις και, και εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτον, εποπτικές εργασίες που συμπεριλαμβάνουν και την Europol και Eurojust. Δεύτερον, συμβουλευτικές εργασίες. Συμβουλεύουμε δηλαδή τον Ευρωπαίο νομοθέτη ε, όταν έχουμε νέες νομοθετικές πράξεις, ε, καθώς και ε, εκτελεστικά μέτρα. Επίσης, ε, παρακολουθούμε τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα πληροφορικής, που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων. Τρίτον, έχουμε συνεργασία, δηλαδή στενή συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, συνήθω γύρω Συνήθως μέσα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, στο οποίο παρέχουμε και γραμματική υποστήριξη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ύπαρξη ανεξάρτητου επόπτη αποτελεί απαραίτητο μέρος της προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως θεσπίζεται και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει λοιπόν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Ο βασικός κανονισμός ε, είναι αρκετά αναλυτικός Και εδώ και δύο δεκαετίες άρχισαν να δημιουργούνται τέτοιοι φορείς. Αναμένεται να συνδυάσουμε τα καθήκοντα του ε, διαμεσολαβητή, ε, του ε, ελεγκτή, συμβούλου, διαπραγματευτή και οργάνου επιβολής του νόμου. Αυτό το μοντέλο βλέπουμε ότι, ότι αντιγράφεται γενικά σε όλο τον κόσμο. Τα γεγονότα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, τον Edward Snowden το 2013, την Cambridge Analytica το 2018, έχουν θέσει τα θέματα προστασίας δεδομένων στο κέντρο της, πολιτικής, της δημόσιας συζήτησης. Πολύ συχνά άνθρωποι λαμβάνουν διαφημίσεις για πράγματα που μόλις αγόρασαν ε, στο διαδίκτυο. Πριν ε, τα τελευταία 20 χρόνια ψηφιοποίηση ε, έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο και πολύπλοκο οικοσύστημα δεδομένων. και οι διάφορες ε, συσκευές ε, γίνονται όλο και πιο διαλειτουργικές μεταξύ τους. Ανησυχούσαμε ότι οι φετινές ευρωπαϊκές εκλογές Ε, θα ήταν η στιγμή που θα άρχισαν να χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για πολιτική χειραγώγηση. Αλλά φαίνεται ότι τα εχέγγυα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν γενικά αποτελεσματικά. Εξετάσαμε πώς το Κοινοβούλιο ε, χρησιμοποιεί τα ε, κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τα προσωπικά δεδομένα για να επικοινωνεί με το κοινό στις προεκλογικές εκστρατείες. Μετά από τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοθεσία πέρσι τον ε, Οκτώβριο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ω επόπτη, έχουμε ε, πραγματοποιήσει 13 επιθεωρήσεις και επισκέψει σε φορεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τελευταίο χρόνο και ήδη φέτο έχουμε οργανώσει περισσότερε καταρτήσει από ό,τι ε, από ό,τι πέρσι. Και μια σημαντική εξέλιξη ήταν ε, η αρμοδιότητά μας να εποπτεύουμε ε, τους τομείς επιβολής του νόμου και δικαστικής συνεργασίας. Από το 2017 εποπτεύουμε την Europol αλλά και την Eurojust αρχίσουμε να εποπτεύουμε φέτος και στο μέλλον θα εποπτεύουμε και τον για ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη είχαμε τέσσερις επιθεωρήσεις της Europol ε, και η επιθεώρησή μας αυτή συμπεριλάμβανε και το πρόγραμμα ε, παρακολούθησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης, Έχουμε ξεκινήσει εξ αποστάσεω επιθεωρήσεις ε, των ιστοσελίδων και των ε, συστημάτων πληροφορική των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Οργανισμών. Ο κανονισμός 2018-1725 ενισχύει τις ε, συμβουλευτικές μας εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας συμβουλεύεται όσον αφορά νομοθετικά μέτρα και συμφωνίες με τρίτες χώρες και ε, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και ο Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ε, ε, μπορούν να γνωμοδοτήσουν και εάν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν μια γρήγορη αντίδραση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Είμαστε στη διάθεσή σας. Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στον τομέα της ε, των τεχνολογιών ε, πληροφορίας ε, και επικοινωνίας είναι κεντρικό μας καθήκον και ξεπερνάει τον απλό συμβουλευτικό μας ρόλο προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σας καλούμε ε, να γίνετε συνδρομητές ε, στις εκθέσεις μας, EDPS Tech Dispatch, που περιγράφουν τεχνολογικές ε, καινοτομίες και αξιολογούν τις συνέπειες για την προστασία των δεδομένων. Στο τελευταίο τεύχος αναφέρουμε του, τα FEE e, ηχεία και τους εικονικούς βοηθούς όπως είναι η Alexa, το Google Home Assistant κλπ μέσα στο πρώτο έτος της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να αναμένουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, τεχνητή νοημοσύνη, που θα έχουν σημαντικές συνέπειες για την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω ότι η χρήση τεχνολογιών ε, τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται ε, αποτελεσματικές νομικές και ηθικές εγγυήσεις. Όταν χρησιμοποιείται η τεχνική νοημοσύνη στην Ευρώπη, θα πρέπει αυτό να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι συζητήσεις με τρίτες χώρες επίσης ε, είναι σημαντικές για μέσα, διότι η προστασία δεδομένων έχει γίνει πια γεωπολιτικό θέμα. Πρέπει να εξετάζονται οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες ε, από τις αρχές προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ενώ παρότι είμαστε μία από τις 29 αρχές προστασίας δεδομένων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, πιστεύουμε ότι είναι μοναδικός ο ρόλος μας. Πιστεύουμε ότι ε, είμαστε η μόνη αρχή που μιλάει με ευρωπαϊκή προοπτική όσον αφορά αυτές τις προκλήσεις και τα όσα πρέπει να κάνουμε στο εγγύς μέλλον. Οι αρχές προστασίας δεδομένων ε, έχουν πια νέα εργαλεία στα χέρια τους. Αυτό θα το δούμε στο εγγύς μέλλον, διότι ε, οι υποθέσεις που αφορούν ε, τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων ε, πρέπει να είναι μετά την 25η Μαΐου 2018. Η επεξεργασία των δεδομένων μας είναι το πιο σημαντικό μας θέμα και πέρα από το φιλόδοξο θεματολόγιο της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες όπως είναι η ε, κανόνες για την προστασία του ιδιωτικού βίου, κάτι που δεν ολοκληρώθηκε κατά την προηγούμενη θητεία. Και που σχετίζεται και με τις διαφορές ε, όσον αφορά την εποπτεία του λεγόμενου τρίτου πυλώνα. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι πάντα ο βασικός μας σύμμαχος όταν αναζητούμε μια κοινή προσέγγιση στα θέματα αυτά. Τέλος, θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς να συμμετάσχετε ε, στην εκδήλωση που οργανώνουμε στη μνήμη του Τζοβάνι Μπουταρέλη που θα πραγματοποιηθεί ε, στις 10 Σεπτεμβρίου στο Concert Noble, 10 ε, λεπτά από εδώ με τα πόδια. Θα λάβετε πληροφορίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εκδήλωση αυτή. Είμαι στη διάθεσή σας και ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο που μου δώσατε. Μου ζητήσατε να μιλάω πιο αργά, γι' αυτό το έκανα. Ευχαριστώ κύριε Βοβ ο Ρόσκι. Το είπα καλύτερα αυτή τη φορά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ε, παθιασμένη παρέμβασή σας. Οι διερμηνείς όμως δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Μιλούσατε πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα είπατε. Καταρχάς να σας πω ότι εχθές ε, τηρήσαμε ενό λεπτού συγγύη για τον κύριο Μπουταρέλη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος ε, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Και το τηρήσαμε προς τιμήν του και ω ένδειξη ε, μνήμη και σεβασμού, διότι ήταν ένας άνθρωπος ε, ε, που έχερε τις εμπιστοσύνη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ένας άνθρωπος προασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών, εμπειρογνώμονα στα θέματα προστασίας δεδομένων, που συνεισέφερε με πάρα πολύ ουσιαστικό τρόπο στην ευαισθητοποίηση για την ε, ανάγκη να προστατεύονται τα δεδομένα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής και όπως είπατε και εσείς και σε δεοντολογικό επίπεδο για την προστασία των δεδομένων, σε ηθικό επίπεδο ε, για την προστασία προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων. Και το αποτύπωμά του δεν ήταν μόνο ευρωπαϊκό, ήταν παγκόσμιο. Γι' αυτό ακριβώ και η διεθνή διάσκεψη που έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ε, δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς τη λαμπρή του ε, οργάνωση. Γι' αυτό ακριβώς, για όλους αυτούς τους λόγους, για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκεστε εσείς εδώ σήμερα και έχουμε και κάποιους ανθρώπους που έχουν ζητήσει το λόγο. Εγώ προσωπικώς ε, που έρχομαι από τον παλιό κόσμο πριν αλλάξει το τεχνολογικό ε, σύστημα και μου στοιχίζει πάρα πολύ να κατανοήσω πάρα πολλά κάποια από τα πράγματα τα οποία αποκτούμε πάρα πολύ γρήγορα ε, που πρέπει να τακτοποιήσουμε, να διοχετεύσουμε, να διαρθρώσουμε, γιατί το γεγονός ότι έχει αλλάξει τεχνολογία δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει η δημοκρατία μας και οι θεμελιώδεις της αξίες. Γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, πολύ συγκεκριμένα ε, αν θέλετε να μα δώσετε κάποια παραπάνω συμβουλή εδώ στην Επιτροπή, η οποία ξεκινάει τώρα, έχει πολλούς νέους βουλευτές. Αν υπάρχει κάτι επιπλέον που θα θέλατε να μας υποδείξετε για τις εκθέσεις τις οποίες θα πρέπει να εκπονήσουμε το επόμενο διάστημα, ακριβώς για το θέμα των δεδομένων και θα δώσω το λόγο πριν ε, να απαντήσετε στον κύριο Μπράιερ, καταρχάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπράιερ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τον οργανισμό σας. Όπως ξέρουμε, το Συμβούλιο θέλει να τον περικόψει κατά πολύ. Ενώ ταυτόχρονα εσείς ε, είστε επιφορτισμένοι με, με περισσότερα. Μπορείτε να μας πείτε πόσες διασυνοριακές ε, ε, υποθέσεις σας απασχολούν ε, την τρέχουσα στιγμή και κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι ο προπολογισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, καλύπτει τουλάχιστον τα ελάχιστα ή αναρκεί τέλο πάντων. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη. Thanks, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και τα συλληπιτήριά μας για ε, τον χαμό του ε, επόπτη. Ήθελα να ρωτήσω για την υπόθεση ΣΡΕΜ, ο οποίος υπέβαλε μια καταγγελία για να σταματήσει η διαβίβαση ε, δεδομένων από το Facebook εκατομμύρια χρηστών από την Ιρλανδία και από άλλες χώρες. Το τεράστιο σκόνδαλο που αποκάλυψε ο Edward αλλά απορρίφθηκε ως απερίσκεπτο βρέθηκε αναγόμενο σε μια υπόθεση που βασιζόταν στη δική του καταγγελία και διατρέχει κίνδυνο να λάβει πρόστιμο εκατομμύριων και η, η ρίζα του προβλήματος είναι ότι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ε, έχουν τα κεντρικά τους στο Δουβλίνο, οπότε ο Ιρλανδός Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων ουσιαστικά ρυθμίζει σε όλη την Ευρώπη τα πάντα για αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς. Ε, η Ιρλανδική κυβέρνηση, όπως φαίνεται, ουσιαστικά ε, κάνει λόμπινγκ για το Facebook και άλλες τέτοιες εταιρείε ε, Και ο παλιότερος πρωθυπουργός Ιρλανδίας κοκορευόταν ότι ήταν καλός φίλος του Facebook και ότι αποδυνάμωνε παλιότερους κανονισμούς και ο, ο, επίτροπος, ο Ιρλανδός Επίτροπος χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Γνωρίζετε όλη αυτή την κατάσταση. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει κάποια άποψη γι' αυτό. Τι θα κάνετε για να υποστηρίξετε την ανεξαρτησία της ε, Ιρλανδικής, του Ιρλανδού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ε, δεδομένης αυτής της τεράστιας επιρροής των ε, πολυεθνικών. Τώρα που έχουμε τον κανονισμό θα ξαναδούμε τέτοιε περιπτώσεις όπως αυτή η υπόθεση Σρέμς. Τι έχετε να πείτε και τέλος γνωρίζετε ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί σε ένα τεράστιο σκάνδαλο για την εισαγωγή της de facto εθνικής ταυτότητας χωρίς καμία νομοθετική βάση. Το γνωρίζετε ή τέτοιου είδου δράσεις θα οδηγήσουν υπό τον κανονισμό σε χρηματικά πρόστιμα, σε χρηματικές κυρώσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Δάλη, ευχαριστούμε. Η κυρία Αλάμοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση των εργασιών του EDPS. Ε, Βασικό στόχος σας είναι να προστατεύετε τα προσωπικά μας δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, για την κατάσταση στην Πολωνία. Όπως γνωρίζετε, ο σημερινός ε, επιθεωρητής αρμόδιος για τα προσωπικά δεδομένα ε, έλαβε αποφάσεις ε, συνέπεια των οποίων το κυρίως γραφείο του Πολωνικού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να, δω, να δημοσιοποιεί πληροφορίες για το ποιους δικαστές, ποιους δικαστές ποιος έχει διορίσει ποιους δικαστές το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί στη ΛΥΜΠΕ. Θεωρείται παραβίαση του νομοθεσία ε, του κράτου δικαίου. Εσεί τι θεωρείτε, Θεωρείτε ότι η απόφαση αυτή ήταν ε, αιτιολογημένη. Ευχαριστούμε κυρία Νταμόβιτς. Το λόγο έχει κυρία Εστσίκ. Εκτός μικροφωνίου μιλήτρια δεν ακούγεται. κυρία Στρίκ και εγώ θέλω να σας δώσω τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο του κυρίου Μπουταρέλη. Πρέπει να είναι τεράστια η απώλεια. Ήμουν μέλος της Γερουσίας της κατοχώρες και εκεί παρατήρησα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο EDPS και για την εθνική νομοθεσία. Ξέρω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα τέτοιο επόπτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο ανταλλάσσει δεδομένα και συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών ε, δεδομένων με τρίτες χώρες και αναρωτιέμαι ο Ευρωπαίος Υπόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει επαρκή μέσα και δυνατότητες να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά στις τρίτες χώρες γιατί αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό αφού υπάρχουν κάποια εχέγγυα μεν, δεν γνωρίζουμε ωστόσο αν τελικά εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό, αν χρησιμοποιείται για άλλου σκοπού. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίπελ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Έχασα την εισαγωγή σας γιατί ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δώσω τα συλληπιτηριά μου για την απώλεια του συναδέλφου Μπουταρέλη για πολλά χρόνια είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και δεν θα είναι εύκολο να συνεχιστεί. Ε, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε πολύ καλή συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα ώστε να μην υπάρξουν και και, ε, και να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τις καλές συμβουλές που λαμβάναμε από τον οργανισμό σας. Ήθελα να κάνω μια, ε, κάποιες ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένε. Είδαμε και μια παρουσίαση της Ευρωπόλ νωρίτερα η συνάδελφό μου το ανέφερε ήδη, όλο και περισσότερο συναντάμε το πρόβλημα συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα δεδομένα που μοιραζόμαστε με αυτές τις τρίτες χώρες. Τι είδου εγγύσεις έχουμε ότι αυτά τα δεδομένα την χάνουν σωστής μεταχείρισης. Το άλλο πρόβλημα φυσικά αντίστροφα είναι ότι αν μπορείτε εσεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να υποστηρίζετε την Ευρωπόλη και τους άλλου οργανισμούς όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα δεδομένα που λαμβάνουμε εμεί, Αντίστροφα δηλαδή και αυτή είναι σημαντική ερώτηση. Επίση, θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση που αφορά τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Σήμερα έχουμε το νέο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συγκεντρώνει όλους τους εθνικούς επόπτες ε, προστασίας δεδομένων Μιλάμε για ένα one-stop shop, για ένα σημείο ενιαία εξυπηρέτηση και σε πολλού τομεί πολλά ερωτήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων που προέρχονται από, τις, ε, από τα 28 κράτη-μέλη καταλήγουν στην Ιρλανδία. Και το λέω γιατί αναφερθήκαμε στο Facebook το οποίο έχει έδρα στην Ιρλανδία. Και διαρωτώ με, έχοντας υπόψη μου τον κανονισμό εργασίας αυτού του Συμβουλίου εσωτερικά, υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν να μην ε, ασχολείται ο Ιρλανδό CDPS με όλα αυτά τα ζητήματα, διότι μπορεί να είναι υπερβολικά πολλή δουλειά για αυτούς. Ε, εγώ ξέρω ότι διεύρυναν το προσωπικό του ο Ιρλανδό επόπτη προστασία δεδομένων, αλλά όχι πολύ. Τι συνεργασία λοιπόν υπάρχει με το Συμβούλιο, υπάρχει κάποια εξέλιξη, πώ εξελίσσονται τα πράγματα, τι γίνεται με κάποια πρώτα αιτήματα που υποβλήθηκαν μετά από την πρακτική υλοποίηση του κανονισμού προστασίας δεδομένων. Έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα. Έχουμε καμιά ιδέα του πώς ε, θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια και αν οι εθνικοί επόπτες προστασίας δεδομένων είναι ήδη επαρκώς εξοπλισμένοι για να κάνουν τη δουλειά τους, να τηρούν τους κανόνες και να ελέγχουν ότι τα πάντα συμμορφώνονται με τους κανόνες του κανονισμού ή εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο περιθώριο λιγμών, για να το πω έτσι, στα κράτη. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Θα ολοκληρώσουμε το γύρο των παρεμβάσεων με την κυρία Νίτβελτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήμουν στο πρώτο μέρος της εισαγωγής σας. Ε, αλλά ήθελα και εγώ να ξεκινήσω δίνοντας τα συλληπιτεριά μου για τον ε, κύριο Μπουταρέλη. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια ε, και είμαι συγκλονισμένη. Λυπήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα για, την απολία του. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, έχουμε ψηφίσει πολλά νομοθετήματα τελευταία, τελευταία χρόνια, το GDPR, και ακόμα μελετάμε διάφορα άλλα. Είμαστε πολύ καλοί στο να νομοθετούμε. Ε, εκεί που χωλένουμε είναι η εφαρμογή. Όλο και περισσότερα ερωτήματα γεννώνται όσον αφορά την ε, υλοποίηση. Έχουν να κάνουν εν μέρη με τα ανεπαρκή μέσα, όπου νομίζω τα κράτη-μέλη ουσιαστικά δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, δεν διαθέτουν επαρκή μέσα στους εθνικούς επόπτες προστασίας δεδομένων, αλλά και το ευρωπαϊκό επίπεδο και τους οργανισμούς επιβολής. Ε, ε, αυτό που με εκπλήσει είναι ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός, βρέθηκαν ε, κάποιες υποθέσεις σοβαρές και επιβλήθηκαν δύο σοβαρά πρόστιμα σε κάποιες εταιρείες ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, στο μεταξύ που δεν φημίζονται για την προστασία των δεδομένων του, επιβάλλουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα. Δεν λέω ότι πρόκειται για κάποιο συναγωνισμό τώρα, αγώνα, ποιο θα επιβάλλει τα καλύτερα πρόστιμα, αλλά πρέπει να το δούμε. Επίση, υπέβαλα ένα αίτημα πρόσβαση ε, στα εγγράφα στο EDPB. Είναι πιθανώ η πρώτη αίτηση τέτοια που έχουν λάβει και θα το γνωρίζετε γιατί Κάτι που δεν λαμβάνουμε υπόψη ε, επαρκώς τα τελευταία χρόνια είναι η διαφάνεια της λήψης αποφάσεων εντός του EDPP και της σχετικής ομάδας εργασίας. Και τέλος ε, θα ήθελα να μου πείτε, αλλά δεν ξέρω αν το είπατε ήδη στις αγωγικές σας παρατηρήσεις, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά πρώτον την, το ηλεκτρονικό απόρριτο αλλά και την αστυνομική οδηγία όπως ονομάζεται που έχει θετηθεί έχει τεθεί σε ισχύ και φαίνεται να την αγνοούν τα κράτη-μέλη. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η αστυνομική οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί με έναν κανονισμό που να προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων από την αστυνομία, το δικαστικό σώμα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών, όπως το GDPR. Ευχαριστώ. Ωραία. ολοκληρώνοντα με τα λόγια της κυρία Σίνεντβελ τις ερωτήσεις ε, και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έκαναν. Κύριε Βιβερόσκη, έχετε 15 λεπτά για να απαντήσετε. Πολύ συγκεκριμένα και ή δυνατόν με τρόπο ώστε οι διερμηνείς να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά του Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής και όσο το δυνατόν πιο αργός. Ε, να μιλήσω για κάτι που ούτως ή άλλως είναι η, επαγγελματική μου σταδιοδρομή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι το οποίο ρωτήθηκα εδώ είναι αν έχω κάποια συμβουλή να δώσω προς τους νομοθέτες. Προφανώς ε, έχω πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες ε, κατά πάσα πιθανότητα είναι τμήμα του έργου του νομοθέτη, αλλά αυτός δεν είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου επόπτη ε, δεδομένο να προτείνει ε, νομοθεσία. Αυτός είναι μόνο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, περιμένω ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το μέλλον θα ασχοληθεί και με τα προβλήματα τα οποία είναι προφανή και που ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε ως ε, κάτι το οποίο αφορούν το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα μας αφορούν ήδη. Και η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι ένα εξαιρετικό ε, παράδειγμα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονική φαντασία και θα συμβεί στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη. Πολλές από τις συσκευέ που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή ήδη χρησιμοποιούν κάτι το οποίο θα μπορούσε να ε, θεωρηθεί τεχνητή νοημοσύνη ή χρησιμοποιούν τα στοιχεία ε, ε, των μηχανών ανάγνωσης, των script ε, μηχανό ανάγνωσης και δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι αλγόριθμοι για τους οποίους θα πρέπει να συζητήσουμε και πώς οι νέοι αλγόριθμοι ε, δημιουργούνται από τους προηγούμενους αλγόριθμους. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Αυτό ακούστηκε και από άλλους που έθεταν τις ερωτήσεις. Υπάρχουν ήδη κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το e-privacy είναι σίγουρα το πιο σημαντικό εξ αυτών, διότι... Ε, ο GDPR ε, με κάποιο τρόπο ήρθε εγκαίρος. Ήμασταν ε, έγκαιροι επίσης, αλλά ίσως και κάπως καθυστερημένοι, για ε, τον κανονισμό προστασίας δεδομένων για τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς θεσμούς και τους οργανισμούς και υπηρεσίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία σε αυτό το μοσαϊκό, τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, αλλά να μην ξεχάσουμε και όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν ή έγιναν εν μέρη στο παρελθόν. Η κυρία Ίνεντφελ στην ερώτηση της ρώτησε και για έναν κανονισμό ο οποίος ε, έγινε στο παρελθόν με ένα, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκεί η οδηγία για το τρίτο πυλώνα. Στην ε, διακοινοβουλευτική συνάντηση ε, Παϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων το 2012 συζητήθηκε το θέμα αυτό και ο Πολωνός Επίτροπος τότε είχε την τιμή να απαντήσει ε, στην ερώτηση σχετικά με την οδηγία και όταν του είπα ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι μπορεί να υπάρχουν και κάποια θεσμικά ζητήματα και συνταγματικά ζητήματα ε, εάν ε, η πράξη αυτή ε, γίνει κανονισμός Εάν όμω έχουμε ένα κανονισμό ο οποίο μοιάζει με οδηγία, γιατί να μην κάνουμε μια οδηγία που θα μοιάζει με κανονισμό. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδίω αυτών που σχετίζονται με τα big data και τις νέες τεχνολογίες ε, για τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι ότι υπάρχει το υπόβεθρο για την εποπτεία όλων αυτών. Ε, υπάρχει αυτό το υπόβαθρο, θα έλεγα, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στους ε, φορείς και στους οργανισμούς και αυτή είναι και η θέση μου ως Ευρωπαίος επόπτης ε, ε, δεδομένων, αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω για το κατά πόσον ισχύει αυτό σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να υπάρχουν λοιπόν κανόνες οι οποίοι είναι περισσότερο σαν κανονισμός είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά πρώτα θα πρέπει να ελέγξουμε αν εφαρμόστηκε η οδηγία στο παρελθόν. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Αν πάρουμε την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ξέρω ότι καταρτίζουν τη σχετική έκθεση για το πού βρίσκεται η εφαρμογή της οδηγίας, μπορεί να απαντήσουμε και στο με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μια ερώτηση για θέματα προπολογισμού. Ξεκινήσαμε με την πρόταση η οποία ε, δόθηκε από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σε γενικές γραμμές ε, την αποδέχθηκε και την προσέθεσε στο Γενικό Προϋπολογισμό, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Επιτροπή. Κατά την άποψή μας, αυτή η πρόταση που δόθηκε εκεί ήταν επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσει που έχει το EDPS για να μπορέσει να κάνει ε, όσα τις αναλογούν και ως τμήμα των θεσμικών οργάνων αλλά και ως συντονιστής και ως γραμματεία του Ευρωπαίου ε, Συμβουλίου ε, Προστασίας Δεδομένων. Έγιναν τεράστιες περικοπές και φυσικά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι η τελευταία κουβέντα στην όλη διαδικασία. Εκτιμήσαμε και τι πόρους λαμβάνουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια στις αρχές προστασίας δεδομένων ε, της κάθε χώρας και διαπιστώσαμε ότι η αλλαγή ήταν περίπου 25% του προϋπολογισμού δηλαδή 25% αύξηση στον προπολογισμό. Και αυτό είναι αυτό το οποίο προτείναμε ε, και μάλιστα να γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν για το 2019 και η δεύτερη για το 2020. Ενώ το πρώτο έγινε και ο προπολογισμό μας για φέτος ε, φαίνεται καλός ε, για τον οργανισμό μας, ελπίζουμε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο όπως συζητήθηκε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από, με την Κομισιόν πριν από ένα χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε έχουμε για τον προπολογισμό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ και να πω ότι η κατάσταση είναι τραγική, αλλά αν θέλει κανεί ε, να έχει αποτελεσματική αρχή προστασία δεδομένων, θεωρώ ότι η πόρη αυτή είναι απαραίτητη. Η επόμενη ερώτηση αφορά την υπόθεση ΣΑΜΣ και την όλη σειρά υποθέσεων που ξεκίνησε ο Μάρξ Ρέμς. Ε, δεν θα ήθελα να πω τι θα γίνει με την παρούσα υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου, γιατί ε, θα ήταν άδικο για μένα να πω τι θα συμβεί. Δεν έχουμε καν ε, την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Ε, θα τη λάβουμε αρχές Δεκεμβρίου. Αλλά θα ήθελα να πω ως κάποιος ο οποίο προέρχεται και από το πανεπιστημιακό τομέα, ότι εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένο για την υπόθεση Μάρξ Ρέμ όταν ξεκίνησε. Πρόκειται για ένα φοιτητή, ο οποίο έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι αρχέ προστασία δεδομένων πριν από 10 χρόνια. Και το λέω ε, ω κάποιο που ήμουν αρχή προστασία δεδομένων. Ο Μάρξ Ρέμ μα είπε ότι, κοιτάξτε, υπάρχουν οι κανόνε και εγώ διδάχτηκα στο πανεπιστήμιο ποιοι είναι οι κανόνε και πραγματικά εσεί δεν ρωτάτε αν έχουν αποτέλεσμα οι κανόνε, αν εφαρμόζονται. Υπ' αυτή την έννοια ε, ικανοποιήθηκα πάρα πολύ για τα όσα έγινα. Είναι δύσκολο όμως για μένα να αξιολογήσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το, ε, οι συνέπειες ε, της υπόθεσης που βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσα τώρα να κάνω σύγκριση μεταξύ της στιγμής που ο Μάρξ Ρέμς ξεκίνησε τον αγώνα του και την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της κατάστασης που είχαμε πριν από την GDPR και την κατάσταση που βιώνουμε τώρα. Ε, όταν ξεκίνησε, σίγουρα, ε, όλοι τα έστελνα στην Ιρλανδία. Και αυτό μπορούσαμε να κάνουμε κι εμεί ω ε, ε δεδομένων. Τώρα που έχει περάσει το GDPR υπάρχει ένα σύστημα ενιαία στηρίδα, υπάρχει το σύστημα της εποπτείας για τα όσα συμβαίνουν ε, στις εθνικές αρκές και παρά το γεγονός ότι ε, ορισμένες φορές κάποιοι διαμαρτύρονται ότι είναι χρονοβόρο και ότι παίρνει πολύ χρόνο, ε, εγώ ε, που συμμετέχω και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού ε, ε, Επόπτη Δεδομένων είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό γιατί η Ιρλανδία μα παρουσιάζει κάθε μήνα τι συμβαίνει στι υποθέσει και το συζητούν οι αρχέ προστασία δεδομένων. Επιτρέψτε να σα πω και κάτι προσωπικό που δεν θα έπρεπε κανονικά να το πω, αλλά ανέκαθεν ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικό όταν άρχισα να δουλεύω στην ομάδα εργασία του άρθρου 29 για την αποτελεσματικότητα καμιά τέτοια ομάδα που απλώ μετράει τον εγωισμό των ανθρώπων που ε, βρίσκονται εκεί. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να καταλήξουν και σε κοινά συμπεράσματα και θα ήθελα να το πω και ως απάντηση στις ερωτήσεις για τις δυνατότητες που έχουν οι Ιρλανδοί συνάδελφοι που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις υποθέσεις. Δεν μπορούμε να τους πάρουμε τις υποθέσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε. Αλλά είμαστε σίγουροι ικανοποιημένοι και είμαστε ανοιχτοί για να τους βοηθήσουμε καθιονδήποτε τρόπο για να μπορέσουν να προχωρήσουν τις υποθέσεις. Ο μηχανισμός συνεργασίας λοιπόν που υπάρχει πραγματικά είναι πολύ αποτελεσματικός. Ms. Ε, κυρία με ρώτησε για την κατάσταση στην Πολωνία. Είναι η μητρική μου γλώσσα η πολωνική. Θα μπορούσα να απαντήσω και στα πολωνικά, αλλά θα απαντήσω στα αγγλικά, γιατί η πρώτη μου απάντηση είναι ότι δεν μπορώ να σχολιάσω την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, στην ε, εθνική δικαιοδοσία και στην κατάσταση των αρχών προστασίας δεδομένων. Είναι κάτι ε, για το οποίο δεν έχουμε εμεί εντολή ω επόπτη δεδομένων και δεν θα έπρεπε να λέω κάτι τέτοιο. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Αν είχαμε ένα αντίστοιχο αίτημα λοιπόν για ενημέρωση για πρόσβαση στα έγγραφα, το οποίο θα το υπέβαλε κάποιο σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα και υπήρχε η απόφαση από το δικαστήριο που έλεγε ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να δοθούν γιατί είναι δημόσια έγγραφα, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η διαφάνεια θα είναι πιο σημαντική αυτή τη στιγμή από την προστασία της προσωπικής ζωής κάποιου και σίγουρα ε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα σε ένα έγγραφο δεν σημαίνει ότι τίθεται θέμα ιδιωτικότητας του εγγράφου και εμπιστευτικότητα του εγγράφου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο Ευρωπαίο Επόπτη θα μπορούσε να αμφισβητήσει την απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά όπω σα είπα, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να συμβεί στην Ευρώπη και δεν αποτελεί σχόλιο στην απόφαση και την ομοθεσία στη χώρα καταγωγή μου. Ε, υπήρξε και μία ερώτηση για την Ευρωπόλ και τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα. Θα θυμάστε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τη διαβίβαση δεδομένων στις 8 χώρες της ε, περιοχής της Μεσογείου, ότι υπάρχει διαφορετική κατάσταση σε κάθε χώρα. Ε, υπάρχουν αυτές οι οποίες δεν έχουν καθόλου κανόνες ιδιωτικότητας και αυτές οι οποίες θεωρούνται ακατάλληλες χώρες βάσει ευρωπαϊκού δικαίου, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ. Ε, το αίτημα για την εντολή ήταν ε, αντίστοιχο για όλες τις χώρες όμως αυτές. Το μόνο που θα μπορούσα να σας πω εδώ είναι ότι προσπαθούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τη Europol ε, σε όλες αυτές τις διαδικασίες προβλέπεται στον κανονισμό της Ευρωπόλ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πιθανής ε, διαβίβασης ε, προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Οκτωβρίου γίνει τρίτη χώρα. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για την Ευρωπόλ και επίσης προετοιμάζουμε και τη συμφωνία πλαίσιο που δημιουργήσαμε με τις τρίτες χώρες ε, για τη διαβίβαση δεδομένων. Ο ρόλος βεβαίως του επόπτη είναι όχι μόνο να ε, συμβουλεύει αλλά και να σταματά κάποιες δραστηριότητες αν δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Ε, και η Ευρωπόλ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη δουλειά. Ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος μου σιγά σιγά. Υπήρξε και μία ερώτηση για την επιβολή. Μπορείτε να μου πείτε τους αριθμούς των υποθέσεων. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ήδη ξεκίνησαν χιλιάδες υποθέσεις ε, ε, στο Συμβούλιο. Έχουμε 616 υποθέσεις διασυνοριακής συνεργασίας που είναι στην βάση δεδομένων του επόπτη, 435 υποθέσεις ξεκίνησαν βάση προσφυγής και οι υπόλοιπες τις ξεκίνησαν οι ίδιες οι αρχές και επίσης 1.716 διαδικασίες που αφορούν αμοιβαία συνδρομή. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ο αριθμός βεβαίως των υποθέσεων είναι πολύ μικρότερος. Μπορείτε να μου δώσετε τον αριθμό. Η κυρία Νέτφελ είπε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του αριθμού των αποφάσεων που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στην Ευρώπη και τις ε, ε, υποθέσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες και τις αποφάσεις των Αμερικάνικων αρχών στον ίδιο τομέα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες από τις αποφάσεις ε, που έγιναν στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι ουσιαστικά ε, συμβιβασμός μεταξύ των επιχειρήσεων και της FTC ε, που ήταν αυτή η οποία προσέφυγε. Ε, μιλάνε φυσικά για πάρα πολλά χρήματα, 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια δολάρια ε, ο διακανονισμός μεταξύ της κυβέρνησης και του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης μία υπόθεση από χθε ή και 5 εκατομμύρια σε μία υπόθεση με το Facebook. Ε, μπορούμε να σας πούμε τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται στην Ευρώπη, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει σχέση ε, με τις αμερικανικές υποθέσεις. Ε, ε, σε γενικές γραμμές όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να θεωρούν ότι τα πρόστιμα είναι κάτι τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην ανάλυση κινδύνου τους και στα εξοδά τους. Ε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το GDPR μας προσφέρει και μία ακόμα δυνατότητα. Η δυνατότητα αυτή ε, μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση ε, συνέργειας μεταξύ παικτών και αρχών που βρίσκονται στην αγορά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα των όσων κάνει το ε, Ευρωπαίος Επόπτης είναι η έρευνα που κάναμε για τους συμβατικούς όρους ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ενός των μεγάλων παικτών στην αγορά λογισμικού. Και αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ 70 αρχών ε, με την ηγεσία του Ευρωπαίου Πόπτη και του Ολλανδικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, το Ολλανδικό Υπουργείο, το οποίο κατάφερε πολύ καλύτερα ε, καλύτερους όρους από τους όρους που είχαν ε, προσφερθεί από τους άλλους στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες και οργανισμούς. Ελπίζουμε ότι τελικά θα μπορέσει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο και τις γενικότερες απαιτήσει ε, που επιβάλλει ο συγκεκριμένος παίκτη σε κάθε θεσμικό όργανο και σε άλλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή αγορά. Δυστυχώς ε, δεν έχω συγκεκριμένες πληροφορίες για τις ταυτότητες στην Ιρλανδία και δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία θα μπορούσαμε εμείς να παρέμβουμε ως Ευρωπαίος Επόπτης Δεδομένων. Ε, θεωρώ ότι το πρόβλημα των εθνικών μητρών είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ε, στην χώρα καταγωγής μου αλλά και στο Βέλγιο υπάρχει ένας αριθμός ταυτότητας ο οποίος δίνεται σε κάθε πολίτη και σε κάθε κάτοικο ε, και έτσι ε, του συνδέει σε διάφορες βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στη χώρα. Στη Γερμανία θα θεωρούνταν κάτι τέτοιο ερωτικό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Όσον αφορά λοιπόν τα διάφορα εθνικά μητρώα είναι τεράστιες οι διαφορές σε κάθε χώρα και εγώ και με την αρμοδιότητά μου ως ε, βοηθός ε, επόπτης των ε, Ευρωπαίων Επόπτη Δεδομένων δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά και αν ξέχασα κάποια ερώτηση σας παρακαλώ μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Ευρωπαίο Επόπτη ανα πάσα στιγμή, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να ε, σας δώσουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στα θέματα ευρωπαϊκής προστασίας δεδομένων. Υπήρχε και μια ερώτηση της κυρίας Σίνεντφελτ για τη διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Συμβολίου Προστασίας Δεδομένων, το θέμα της επιστολής που μας εστάλει και το αίτημα ε, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βιβερόσκη και με αυτό ευχαριστώντας και τους ευρωβουλευτές, τις ομάδες τους, τους διαρμηνείς και όλους τους παρισταμένους Ολοκληρώθηκα αυτή η πολύ έντονη συνεδρίαση. Νομίζω ότι μας αξίζει ολονών ξεκούραση και αν για σας ξεκούρασε ξεκινάει τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.